So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σήμερα το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σεμινάριό μας με βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων Οργανώσαμε αυτό το σεμινάριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και ε, ξέρετε τα αποτελέσματα των συζητήσεων στα διάφορα φόρα δεν συγκλίνουν πάντοτε. Θα ήθελα ε, να καλωσορίσω επίσης ε, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την κυρία Ρέντινγκ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είστε αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον καθηγητή Σιμεωνίδη, που εκπροσωπεί την Κυπριακή Προεδρία. Να καλωσορίσω την κυρία Νταϊάννα Γόλης, τέος Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι συνεισηγήτρια για το, πρόταση για το ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Δεν θα, θα ήθελα να καλωσορίσω τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να καλωσορίσω και τον Λόρδο Μπόουνες που θα προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ μετά από τις εισαγωγικές παρουσιάσεις. Ε, θα ήθελα να προσθέσω δε και μια παρατήρηση για να σε εκθέσω την προσωπική μου άποψη. Το αποδίδει ιδιαίτερη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αυτό το ζήτημα. Ζητήσαμε και τελικά πετύχαμε ευρύτατη πλειοψηφία για την έκθεση Wallis στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πρόταση που κατέθεσε. Η πρόταση αυτή έχει συζητηθεί επί μακρόν σε διάφορες επιτροπές. Εμείς θα συζητήσουμε το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και όλα τα συναφή ε, με την πρόταση ζητήματα. Το ότι μας εδόθη η ευκαιρία να διοργανώσουμε το σημερινό σεμινάριο καταδεικνύει τη σημασία που έχει το ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, συνιστά μεγάλη πρόοδο για την εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια πρόταση αν τελικά ε, καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία. Θα ξεκινήσει έτσι η ευρωπαϊκή αυτή διαδικασία. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέντιν και στη συνέχεια στον καθηγητή Σιμεωνίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε δίκιο. Αυτή η πρόταση έχει μία ε, μακρύτατη ιστορία, δεκαετιών θα έλεγα. η καλύτερη δικηγόρη μας για το συμβατικό δίκαιο ε, έχουν ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το ζήτημα, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούμε να προσδώσουμε την πλέον κατάλληλη νομική μορφή σε αυτήν την πρόταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε, είναι πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και συνεισηγητής για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γόλισε για την προσήλωση που έχει δείξει για την προώθηση αυτού του ζητήματος και να ευχαριστήσω και τον καθηγητή Σιμεωνίδη, χάρη σε εκείνον η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε επίσης επισταμένα για ε, να προωθήσει αυτό το φάκελο. Ε, μέσα σε αυτή την πρόταση βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη το δικαστικό μας σύστημα. Αυτή η νέα πρόταση θα ρίξει τους φραγμούς που συνδέονται με τα συμβατικά δίκαια, εθνικά συμβατικά δίκαια. Επίσης θα μειώσει το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή διαφορετικών δικαίων, κόστος δυσανάλογα μεγάλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κυρίω. κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Χάρη στην πρόταση θα θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα έχουν ε, την επιλογή να επιλέξουν αυτό το δίκαιο για τις διασυνοριακές συναλλαγές τους ε, ανεξαρτήτως της έδρας των επιχειρήσεων ή του τόπου διαμονής των φυσικών προσώπων θα ενισχύσει επιπλέον την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε σχέση με, την, ε, με το σημερινό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε σχέση με τα εθνικά δίκαια θα αποτελέσει πλεονέκτημα ε, ε, σε όφελος των καταναλωτών διότι θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα με χαμηλότερη τιμή. Είμαι αρμόδια για τα θέματα δικαιοσύνης ε, και βρίσκομαι τώρα ενώπιον των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία και εντάσσονται σε όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κατευθυντήριες γραμμές 10 κατά την κατάρτιση της νέας πρότασης για το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα των πολίσεων σέβονται απολύτω αυτές τις αρχές και γι' αυτό επιλέγουμε εξ αρχής ένα προαιρετικό καθεστώς αντί να ακολουθήσουμε τη συνήθι νομοθετική οδό της πλήρους εναρμόνισης. Ε, δεν αντικαθιστούμε δηλαδή τα ισχύοντα εθνικά συμβατικά δίκαια. Ε, προτείνουμε ένα εναλλακτικό σετ κανόνων ε, διαθέσιμο σε όλα τα εθνικά νομικά συστήματα με τρόπο ώστε οι διασυνοριακές συναλλαγές να είναι ευκολότερες και φθηνότερες ε, ούτως ώστε να γίνονται κάποιε συναλλαγές που αλλιώ δεν θα συνέβαιναν, όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι στοχευμένη δε η πρόταση και καλύπτει μίσο όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα και δεν ε, υπερβαίνουμε αυτά που είναι απαραίτητα για να υπερπηδήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα εμπόδια. Καλύπτει τις διασυνοριακέ συμβάσει και μόνο και όχι ε, συμβάσει ανάμεσα σε μεγάλες επιχειρήσεις για τις συμβάσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις B2B. Ε, συνειδητοποιούμε ότι πρέπει για να εφαρμοστεί το δίκαιο ε, να είναι η επιχείρηση μικροεπιχείρηση ή μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό σε, κατά τη διαστολή με αυτά που ισχύουν ε, βάσει των εθνικών δίκαιων. Ο προαιρετικό χαρακτήρα της πρόταση συνάδει με την αρχή της σύναψης συμβάσεων. Ε, οι, εμπορευόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με τα εθνικά δίκαια έχουν την ε, επιλογή, μπορούν ε, να προκρίνουν το εθνικό δίκαιο αντίθετα. Όσοι βλέπουν τα ωφέλη που συνεπάγεται το εναρμονισμένο σετ κανόνων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εναλλακτική λύση. Είναι δική τους επιλογή. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ένα κοινό ευρωπαϊκό συμβατικό δίκαιο. Είτε πρόκειται για επιχείρηση, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Είναι όμως μια επιπρόσθετη εναλλακτική λύση για όσους την επιλέξουν. Προτείνοντας ε, με αυτή την προαιρετική λύση για το Ευρωπαϊκό Συμβατικό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πλήρη ε, επίγνωση της ε, δυσκολίας ε, που, των δυσκολιών μάλλον ε, που συνεπάγεται η καινοτομία σε αυτόν τον τομέα ε, και συνειδητοποιεί πλήρως ε, το μέγεθο των προβλημάτων και των φραγμών που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Οι συζητήσει τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας ακολουθούν την σωστή κατεύθυνση. Εξετάζονται τώρα και στα δύο θεσμικά όργανα οι διατάξει διατάξεις της νέας νομοθετικής πρότασης ε, και χαίρομαι που διοργανώνονται διάφορα εργαστήρια για να εξεταστούν οι λεπτομέρειες ε, του νέου ευρωπαϊκού δικαίου και μένω τις εκθέσεις από τις διάφορες ομάδες εργασίας ε, από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς τα προσεχή χρόνια ούτως ώστε να διαπιστώσουμε βάσει των κοινών μας προσπαθειών ποια είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Για τα ένδικα μέσα ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί για τη νέα πρόταση από πολιτικής και από οικονομικής ε, σκοπιάς όλοι ενδιαφερόμενοι Εξάλλου, ε, το έχουν αναφέρει αυτό στις δηλώσεις τους. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, αρχικά εξέτασε αυτά τα κεφάλαια και τόνισε την ε, καταλητική σημασία αυτών των πρακτικών ρυθμίσεων. Την ίδια προσέγγιση ιδέα ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέλουν να μεριμνήσουν τόσο ώστε το τελικό κείμενο να χαρακτηρίζεται από την ευέλτιστη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στις νέες δυνατότητες ε, για τις επιχειρήσεις αφενός και τις νέες δυνατότητες για τους καταναλωτές αφετέρου. Η νομική ασφάλεια που χρειάζονται και οι δύο και η απαιτούμενη ευελιξία ούτως ώστε η επιλογή τους να είναι μια πραγματική επιλογή. Ε, και οι δύο συνομοθέτες ε, θα είναι στο πλευρό τους για να κάνουν τι απαιτούμενε αλλαγές, αλλαγές που θα κρίνουν απαραίτητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμμετέχουμε και σε διαλόγους που γίνονται σε εθνικό επίπεδο ε, και επιθυμούμε στις επικείμενες διαπραγματεύσεις να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το νέο νομοθέτημα έχει κάποια θέλγητρα και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που ε, εν καιρό κρίσης θα πρέπει να διευρύνουν τις νέες ευκαιρίες και να χρησιμοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς κάτι που συνιστά ουσιαστική δυνατότητα ανάκαμψης αν καταφέρουμε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της αγοράς να τους φραγμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Ρέντεν, κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στον κύριο Σιμά Σιμανίδη. Ελπίζω πρόφερα σωστά το όνομά σας ε, για την Κυπριακή Προεδρία. Θα λάβει τον λόγο. Έχει τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Σας... ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να με εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, μικρή βέβαια, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Πολιτική της Κυπριακής Προεδρίας είναι να προωθεί κάθε ζήτημα ξεχωριστά και το ξέρω αυτό γιατί εμπλέκομαι εγώ σε όλα τα επιμέρου ζητήματα με τα οποία ασχολείται η Κυπριακή Προεδρία και αυτό γίνεται πάντα ανεξάρτητα από την θέση που μπορεί να έχει κάποιο κράτος μέλος για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ σημαντική πρόοδο σε δύο προτινόμενες ε, νομοθεσίες όσον αφορά τις συμβάσεις συμβίωσης, μολονότι η κυπριακή νομοθεσία δεν αναγνωρίζει τις συμβάσεις αυτές συμβίωσης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα η Κορεπέρα αποφάσισε να προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει συγκεκριμένε πολιτικές κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, δεν κάναμε επιλογή μόνο των σημείων που μας άρεσαν, ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη ενιαία πολιτική, όπως ακριβώς κάνουμε και σε πολλά άλλα ζητήματα. Αυτό ακριβώς κάναμε και το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Προκειμένου να αρχίσουμε να συζητούμε όμως τώρα την ουσία της νομοθεσίας αυτής, θα πρέπει να γίνουν πρώτα κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τους τελευταίους 8 μήνες οι σχετικές ομάδες εργασίες συζήτησαν κάποια προκαταρκτικά ζητήματα, τα οποία όμως είναι εξίσου σημαντικά, όπως για παράδειγμα η νομική βάση και το καθεξής. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουμε να συζητήσουμε την ουσία του ζητήματος αυτού, το ότι καταφέρουμε μάλλον να μπούμε στην ουσία του ζητήματος αυτού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου. Θέλουμε πραγματικά να περάσουμε στα ουσιώδη σημεία και γι' αυτό το λόγο κάναμε κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε αντί να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις από το πρώτο τμήμα του παραρτήματος, ξεκινήσαμε από το τέταρτο τμήμα που περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλωμένων μερών, καθώς επίσης και όλα τα διορθωτικά μέτρα και τα ένομα μέτρα τα οποία διαθέτουν και οι δύο πλευρές. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το σημείο 4, γιατί ακριβώς εκεί πέρα βρίσκονται οι πιο σημαντικοί κανόνες, αυτοί που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό άλλωστε έχει φανεί ιδιαίτερα από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη. Θεωρήσαμε ότι το τέταρτο λοιπόν τμήμα του παραρτήματος θα μας δώσει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την πρόταση αυτή με το κοινοτικό κεκτημένο και με τις εθνικές νομοθεσίες στα κράτη-μέλη. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μια τέτοια συζήτηση και τον να εξοικειωθούμε κάπως με τα ζητήματα τα οποία προτείνονται αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε κάποιου ενδιασμού οι οποίοι είχαν προκύψει. Σαφώ όμω υπάρχουν κάποιε διαφωνίε ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την πρόταση αυτή. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι διαφωνίε αυτέ έχουν κάνει με την ιδέα αν πραγματικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων ή όχι. Εμεί, ω Προεδρία θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μία στάση επικοδομητική ουδετερότητα. Προφανώ οι αποκλήσει αυτέ μεταξύ των κρατών μελών θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον. Θα ήθελα όμω να κάνω και μία προσωπική παρατήρηση βάσει τη ε, εμπειρία που έχω από την ε, ε, διδασκαλία που έχω διεξάγει τα τελευταία 34 χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει και στον τομέα αυτό και οι δύο πλευρές να δείξουν μια θετική στάση. Στην δεκαετία του 1940 κάποιοι σημαντικοί νομομαθείς είπανε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ομοιόμορφος κώδικας εμπορικός. Την εποχή εκείνη οι περισσότεροι είχαν πει ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ένας τέτοιος κώδικας και πολλοί είχαν πει ότι δεν ήταν καν ευκταίος. Πέρα από την γενικότερη αντίδραση που υπάρχει όσον αφορά την κωδικοποίηση του τομέα αυτού σε νομοθεσία. Το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν ότι η εμπορική νομοθεσία των πολιτιών, των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε ποτέ να εναρμονιστεί, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές διαφορές και ότι δεν θα μπορούσε ποτέ εκ των άνων να επιβληθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβληθεί μια τέτοια εναρμονισμένη νομοθεσία, αλλά ότι θα εξαρτιόταν πάντα από την θέληση των διαφορετικών πολιτιών να εφαρμόσουν μια τέτοια νομοθεσία. Οι περισσότερε λοιπόν πολιτείε των ΗΠΑ θεώρησαν δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί ένα τέτοιο εναρμονισμένο εμπορικό κώδικα. Και τελικά όμω πραγματοποιήθηκε μέσα σε δύο δεκαετίε όλε οι πολιτείε των ΗΠΑ είχαν εγκρίνει έναν ομοιόμορφο εμπορικό κώδικα. Οι τελευταίε μάλιστα πολιτείε ενέκριναν τον κώδικα αυτό στα τέλη τη δεκαετία του 70. Θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω να σκεφτείτε κι εσεί μακροπρόθεσμα, επικοδομητικά, με τον ίδιο τρόπο. Να μην ατενίσετε του επόμενου μήνε αλλά τα επόμενα χρόνια, αν θέλετε. Ενδεχομένω να διαφωνούμε για κάποιε λεπτομέρειε του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων και πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε προκειμένου να επερκεράσουμε τι διαφορέ μα και να καταφέρουμε να βελτιώσουμε κάποια σημεία στα οποία η πρόταση αυτή χωλαίνει. Πιστεύω πάντω ότι η εναρμόνιση, αν μη τι άλλο η προσέγγιση των ανοχικών δικαίων των κρατών μελών είναι ένα πολύ καλό στόχο για το μέλλον και στην περίπτωση αυτή το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μπορεί να αποτελέσει ένα καταπληκτικό μέσο προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή τη σύγκληση. Αν τελικά το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων στεφθεί με επιτυχία, τότε όλοι μα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε την επιτυχία αυτή. Και αν πραγματικά ε, το προϊόν αυτό, να θέλετε, είναι καλό, είναι θετικό, τότε θα το ενστερνιστούν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και όλα τα κράτη-μέλη και κάποια στιγμή τελικά μπορεί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν την νομοθεσία αυτή ως εσωτερική εθνική νομοθεσία. Θα γίνει πραγματικότητα λοιπόν τότε το κοινό αυτό ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο δεν θα επιβάλλεται απλώς εκ των άνω, αλλά θα είναι ένα δίκαιο το οποίο οριζόντια θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη με ε, την οικία βούληση των κρατών μελών, επειδή τα ίδια τα κρατη θα το έχουν επιλέξει. Ενδεχομένω να φαίνεται πάρα πολύ μακριά η μέρα αυτή σήμερα, αλλά δεν υπάρχει λόγο να απελπιζόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με το θετικό αυτό τρόπο, να σε ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σα και να ευχηθώ στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία κάθε επιτυχία για το σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Νταϊάννα Γουόλης, επόμενη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ για το ότι με προσκαλέσατε να προσέλθω σε αυτή τη σημαντική συνάντηση για τη συζήτηση για τον, το κοινό Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι κέρια σημασία για να θα ε, κάνουμε σωστά τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ενθαρρυντικό να ακούει κανείς ε, διάφορες απόψεις με παρεμβάσεις επί της ουσίας και όχι λέγοντας αν και σε περίπτωση που και τα λοιπά υπόρους και προϋποθέσεις. Ας ξεκινήσουμε με το αν και τις προϋποθέσεις αυτές, προσεγγίζοντας κάπως διαφορετικά τα πρακτικά μέτρα που βρίσκονται γύρω από αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε στο αν και γιατί. Είναι κάπως και προσωπικό το θέμα αυτό, διότι αυτή η πρόταση αφέ ε, με τις διάφορες ε, πτυχές της με συνόδευε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού μου βίου επί 12 Και έτσι έχει μεγάλη περίοδο κυοφορίας ή γενέσεως, αν επιτρέπεται η έκφραση, αλλά και πέρα από αυτό, για μένα προσωπικά έχει και παλαιότερη προηγούμενη ιστορία. Όταν πριν από αυτή τη δωδεκαετή περίοδο ήμουν ασκούμενη νέα δικηγόρος στο Λονδίνο και όλο το χρόνο μου ως ασκούμενη δικηγόρος ασχολήθηκα με διασυνοριακές διεκδικήσεις και απαιτήσει και είδα από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που ενέχει το θέμα για τα εμπλεκόμενα μέρη που προσπαθούν να συναλλάσσονται διασυνοριακά στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μετά ήρθα εδώ στην Ευρωβουλή και είπα και είδα ότι εδώ επιτέλους μπορούμε κάτι να κάνουμε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να καταστεί πιο εύκολο και πιο ασφαλές η ενιαία εσωτερική αγορά να αποκτήσει σάρκα και οστά και να γίνει πραγματικότητα για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε βέβαια αλλά θα έπρεπε να γίνει και αυτό το τελευταίο βήμα για να καλύψουμε την απόσταση και να καταφέρουμε αυτό το οποίο όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια προαγωγή, μια προώθηση για την ανάπτυξη σε ένα δίκαιο πλαίσιο και πιστεύω ότι και ως δικηγόρος αλλά και ως εκπρόσωπος κοινοβουλευτική, ως βουλευτής, πιστεύω ότι αυτό που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε και να στήσουμε στα πόδια του δεν είναι απλώς κάτι τυπικό που θα αφορά τις ε, αντιπαραθέσεις και τριβές. Είναι κάτι το οποίο είναι προληπτικό στη φύση του, προληπτική νομοθεσία, προληπτικό δίκαιο που θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους ε, καταναλωτές, μικρομεσαίους καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο σε αφετηρία απόλυτα ο ένας τον άλλον στην πρώτη φάση τον του συσχετισμού τους ε, με τους άλλους της απέναντι όχθης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προληπτικά να δράσουμε, να μην καταλήγουμε ε, έχοντας υπόψη ένα στόχο δαπανηρής όλας ε, επιδιατησίας και συμφιλίωσης αφού θα έχει γίνει η ζημιά, αλλά να μπορούμε προληπτικά στις διασυνορικές συναλλαγές να βοηθήσουμε να αποκομίσουν τα μέγιστα ωφέλη οι εμπλεκόμενοι. Περί αυτού θα έπρεπε λοιπόν να πρόκειται και να είναι δεν είναι ένα, ας το πω έτσι, μια κονίστρα, ένα γήπεδο όπου θα υπήρχαν, υπήρχε περιθώριο να δρούν ε, ε, στο παιχνίδι αυτό δικηγόροι επιδιαιτησίας. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε παράλληλα με την συνένεση για το εμπορικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο ε, για να προχωρήσουμε. Κάποιοι θα έλεγαν ότι αυτά τα άλλα στοιχεία είναι πιο σημαντικά κιόλα από το ΚΕΕΔ, το Κοινό Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο. Μπορούμε να συζητήσουμε για παράδειγμα για τη γλώσσα, για την ε, ε, προσέγγιση αυτή. Όμως όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει άρρηκτα να αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων που θα υιοθετήσουμε αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μικρές επιχειρήσεις στην εκλογική μου περιφέρεια μου έλεγαν ότι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και θα είναι πραγματικότητα για μας αν έχουμε όρους και προϋποθέσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας χειροπιαστά, που θα είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία σε όλες τις γλώσσες ε, της ευρωπαϊκής κοινότητας. Και αυτή είναι η ομορφιά, το κάλος της Ευρώπης. Μπορούμε να το κάνουμε και θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε όλες αυτές τις γλώσσες, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις. Θα πάρει πολλή δουλειά, θα είναι εργόδηση η προσπάθεια, κοπιώδηση για να καταλήξουμε στο βέλτιστο προϊόν, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει εύθετα εύθετα η εσωτερική αγορά. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή, ορθή πρόταση. Κατά την κατάλληλη χρονική στιγμή και συγκυρία. Είναι η ορθή πρόταση για δύο λόγου. Διτά, που ήδη προαναφέρθηκαν, σέβεται απόλυτα την αρχή τη επικουρικότητα. Ποιο καλύτερο παράδειγμα επικουρικότητα μπορεί να έχει κανεί και να δει από εσά και εμένα άτομα και εμπλεκόμενους που μπορούν ατομικά να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν κάτι ή όχι. Προαιρετικά, ελευθερία συμβατική, θεμελιώδης αρχή της επικουρικότητας. Και αν όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, θα βοηθήσουν τις οικονομίες μας σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη συγκυρία, μιας πολύ δυσχερούς περίοδου που διανύουμε. Και μια τελευταία σκέψη από πλευράς μου, αν επιτρέπετε. Ως συνεισηγήτρια κατά τους τελευταίους μήνες εδώ στο Κοινοβούλιο, Κάποια στιγμή είχα ένα, μια επίσκεψη, επίσκεψη από την Κίνα. Εξέχων καθηγητής ε, δικαίου και δικαστής Κινέζος με επισκέφθηκε. Περί τίνος ήθελε να μου μιλήσει, ήθελε να αναφέρει το κοινό ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο. Και είναι πράγματι ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι. Εξαιρετικό είναι, υπέροχο αυτό το οποίο κάνουμε εδώ. Και έχω, φοβούμαι ότι αν δεν έχουμε το θάρρος, εμείς άλλοι θα έχουν το θάρρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ, Diana Wallis. Και περνάμε τώρα στο πρώτο πάνελ, στον πρώτο γύρο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Λόρδο Μπόνες. Είναι ο πρόεδρος, προεδρεύων της Επιτροπής για το Δίκαιο και την Προστασία Καταναλωτών της Κάτω Βουλής, υποεπιτροπής στο ε, ε, ε, Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Κάτω Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτός θα αναλάβει τώρα την Προεδρία. Έχετε τον λόγο, Λόρδε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος ε, στις παρατηρήσεις μου, τόσο ώστε οι διακεκριμένοι ομιλητέ που έχουν αναγραφεί στην ημερή σε διάταξη να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς Πρόεδρε και την Επιτροπή σας που συγκάλεσαν τη σημερινή συνεδρίαση και για την πρόσκληση που απίφθηνα σε βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όπως ήδη είπαμε πρόκειται για μια ε, πρόταση με μια πολύ μακρά ιστορία ε, που με στόχο τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν και υπεστηρίζουν ε, τους στόχους της πρότασης αυτής, δηλαδή ενίσχυση της ενίας αγοράς τονώνοντας το στο εμπόριο. Είναι λυπηρό όμω και εδώ αρχίζουν να δει τα απόψεις μιλώντα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως όχι γενικά, αλλά ε, ε, είναι χαρακτηριστικό όπως συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν διάφορα παράδοξα πράγματα, αρκετά περίεργα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όντως δείχνουν ενθουσιασμό, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις όχι τόσο. Ε, τα συμφέροντα των ε, καταναλωτών ε, παραδόξως πως είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή ανησυχούν από διάφορες πλευρές, θεωρούν ότι αυτό το νέο νομοθέτημα δεν θα παράσχει επαρκή προστασία και ενδεχομένω να δημιουργήσει και ασφάλεια. Όμως αυτό αποκλείεται βάσει της πρότασης επίσης ενώ δεν υπάρχουν υποψίες σχετικά με τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πιστήρια, τα τεκμήρια βάσει των οποίων ε, ναι, θα αποδεικνυόταν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των διασυνοριακών συναλλαγών δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και καταλητικά. Οπότε ίσως ε, θα έπρεπε, λένε κάποιοι, να περιμένουμε τη διεξαγωγή μελετών προτού προχωρήσουμε περισσότερο. Υπάρχει βεβαίω και το θέμα της νομικής ε, βάσης. Όλα αυτά είναι ζητήματα μείζων σημασίας. Ε, θα πρέπει να, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα προσεγγίζουμε για να δούμε αν με αντικειμενικό και επικοδομητικό τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή μας, τον διακεκριμένο Σερ Τζον Τόμας, πρόεδρο του σχετικού τμήματος ε, της του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου και σας μιλώ με την ιδιότητα του Προέδρου της ε, σχετικής ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου, όπου ε, ακαδημαϊκοί δικαστές ε, και ενεργεία δικηγόροι εκπροσωπούνται. Το θέμα δεν είναι πολιτικό. Έχουμε κάνει ήδη τις πολιτικές επιλογές ε, και αυτό φάνηκε από ε, και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα αυτού του νέου νομικού μέσου. Πρέπει να είναι καλό αυτό το νομικό μέσο καθότι είναι προαιρετικό διότι θα πρέπει να ανταγωνιστεί με τα όσα ισχύουν σε άλλα νομικά συστήματα και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Θα πρέπει να είναι ε, σαφέστερο, συνεκτικότερο και ασφαλέστερο το νέο νομοθέτημα ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή του. 300 σελίδες είναι η έκθεση που προέκυψε από την ομάδα εργασίας μας. Η δική μου σημερινή πρόκληση είναι σε λιγότερο από 10 λεπτά να τα συνοψίσω όλα αυτά. 10 σημεία λοιπόν. Ε, με μάλλον μεγάλη ταχύτητα για να σας δείξω, να, ε, να αποδείξω αυτά που είπα. Πρώτο σημείο, ε, σε τεχνική βάση υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να απλουστεύσουμε τη δομή του νομοθετήματος. Φερρυπίν, μπορούμε να συντομεύσουμε τους ορισμούς για να εντάσσονται καλύτερα στον κύκλο ζωής της κάθε σύμβασης, να προσδιορίσουμε επακριβέστερα την ορολογία. Δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρέπει να είναι ελκυστική η νέα πρώτη. Δεύτερο σημείο, ε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να απλουστεύσουμε και το πεδίο εφαρμογή. Παραδείγματο χάρη, νέα πρόταση θα έπρεπε να καλύπτει και συμβάσει σε μεικτού μεικτού στόχου, δηλαδή πέρα από τις ε, πωλήσει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ξέρετε ότι στην πραγματική ζωή υπάρχουν και συναφείς υπηρεσίες και δεν περιοριζόμαστε στην ξεκάθαρη συναλλαγή πώληση ενός προϊόντος. Τρίτο στοιχείο, θα έχουμε το ψηφιακό περιεχόμενο, ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή και πρέπει να προσαρμόσουμε τη νέα πρόταση. Οπότε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές ε, στη νέα πρόταση και πιστεύουμε ότι δεν έχει αποδοθεί ιδέουσα σημασία σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Παραδείγματο χάρη η υποχρέωση παράδοση σε βάση της οποίας ε, πρέπει να γίνει η παράδοση του αγαθού, το οποίο δεν έχει νόημα εφόσον μπορεί να πρόκειται για ψηφιακά αγαθά. Τέταρτον, τα συνοδευτικά μέτρα της πρότασης. Ε, θα ακούσουμε και στη συνέχεια κάποια σχετικά πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να ε, ε, εξηγήσουμε καλύτερα το στόχο μιας εναρμονισμένης προσέγγισης. Σε σχέση με αυτά που μας είπε νωρίτερα η κυρία Γουάλης, ε, δεν πρέπει να βγάζουν περισσότερα λεφτά οι δικηγόροι από την επίλυση διαφορών και τους διακανονισμούς. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Θα δούμε αν με τις νέες ρυθμίσεις ή με μια νέα συμβουλευτική επιτροπή με άλλα διεθνή μέσα, με βάση δεδομένων δεδομένων, ένα νέο μηχανισμό για την επίλυση διαφορών. ίσω έτσι μπορούμε να αποφύγουμε ε, το επιπρόσθετο κόστο. Αυτά είναι τα τέσσερα γενικά σημεία. Πέμπτο σημείο. Το πέμπτο σημείο, υπό το πρίσμα των καταναλωτών. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός opt-in εθελοντική συμμετοχή και αρκε, αρκετοί περί, συμμερίζονται την άποψη είναι αρκετά περίπλοκο ε, και πολλά μπορούν να γίνουν να πλουστευτεί αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει η πρόταση ενθαρρύνοντα καταναλωτέ να χρησιμοποιούν αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση σε μια ιστοσελίδα λαμβάνοντα υπόψη ε, τις ε, διατάξεις για την, ε, να επισημαίνεται αυτό. Το Επόμενο σημείο θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε όλες τις ελεύθερε συμβάσει και συμβόλαια για μέσω των διαπραγματεύσεων. Το σημερινό σχέδιο προβλέπει ότι αναδρομικά θα εφαρμόζεται αν συνάπτεται σύμβαση υπό αυτό το καθεστώς. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα ότι δεν θα μπορούσε μέσα στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος να εντάσσεται κάποιος και γι' αυτό θα πρέπει πληροφορίες ε, να διατίθενται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Δεν έχει νόημα εξετάζοντας ένα, ε, το πλαίσιο ενός δικαίου να εφαρμόζεται όταν θα υπάρχει η ανάγκη ο πολιτής ε, να αντιμετωπίζει δύο διαφορετικά ε, νομικά καθεστώτα. Επίσης, ε, η ανάγκη να προσαρμόζεται αυτό το καθεστώς στην ψηφιακή εποχή, με την ανάγκη να υπάρχει μια δυνατότητα προαιρετικής προστασίας πληρωμής. Αν κάποιος αγοράζει ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, θα επιθυμεί να γνωρίζει ότι τα χρήματα τα οποία εμβάζει θα προστατεύονται. Η πληρωμή θα προστατεύεται. Σε περίπτωση μη παράδοσης ε, των αγαθών, των εμπορευμάτων. Προτείνουμε λοιπόν ένα μηχανισμό για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Επίσης ε, κάτι θα πρέπει να γίνει για να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών θα εξισορροπούνται με το σωστό τρόπο σε σχέση με την νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Παράδειγμα, υπάρχουν πολλές περιπτώσει. Ε, όπου η άποψη που θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα δικαστήριο και η επιρροή αυτής της ατομικής άποψης ε, περί του τι εστί καλή προαίρεση και καλές προθέσεις και ισοδίκαιο πλαίσιο συναλλαγής. Θα πρέπει εδώ όμως να δούμε να μην υπάρξει ένα, ένα σχετικός βαθμός νομικής αβεβαιότητας. Είναι λοιπόν πραγματικά σημαντικό να άρουμε στο μέγιστο δυνατό τη νομική αβεβαιότητα ή ανασφάλεια. Μετά ένα το σημείο, ένα την παρατήρηση. Και αυτό τώρα θέλω, θέλω με αυτό να δώσω δύο παραδείγματα σε σχέση με τις συμβάσεις επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις. Το σχέδιο θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε η μερική επιλογή να μπορεί να καλύπτεται. Θα πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι αν επιλέγει αυτό μια επιχείρηση δεν μπορεί η υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων να ε, υπεκφεύγεται. Και τελευταίο σημείο με το οποίο ολοκληρώνω τη σύντομη παρέμβασή μου. Οι θετικές προθέσεις, ε, ε, το θετικό πνεύμα ε, είναι αναγκαία προϋπόθεση. Βλέπουμε το ότι πρέπει εδώ να δούμε την σημασία των όρων και προϋποθέσεων έναντι της, ε, ε, των καλών προθέσεων ώστε να μην υπάρξει ανεξέλεγκτο πλαίσιο. Μία πρόταση που υποβάλλουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει για παράδειγμα ε, αποζημίωση αν παραβαίνει κάποιος αυτόν τον κανόνα. Αυτά συνοψίζοντας μέσα σε 10 λεπτά όλα αυτά τα θέματα με αυτές τις 10 παρατηρήσεις προσπάθησα να δώσω ένα παράδειγμα πώς εμείς θέλουμε με θετική προσέγγιση να ε, είμαστε αρρωγοί και να συνδράμουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τεχνικής, ε, τεχνικού χαρακτήρα θέματα από νομικής πλευράς. Υποβάλαμε μια εναλλακτική ολόκληρη σειρά προτάσεων, διότι θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις ε, χωρίς να βλέπουμε ποιες επιπτώσεις και ποια διατύπωση θα επιλέγεται. Δεν είναι η πρόταση εναλλακτική αυτή, αλλά προτείνουμε απλά αυτά τα οποία εμείς θεωρήσαμε από την επισκόπηση και εξέταση αυτού του μέσου εκείνα τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν στην πρακτική εφαρμογή καλύτερα. Είναι στη δική σας διακριτική ευχαίρεια, Πρόεδρε και στους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να επιλέξετε. Στενερά πιστεύουμε ότι πολλά μπορούν να γίνουν και ελπίζουμε ότι οι επικρίσεις θα είναι επικοδομητικού χαρακτήρα επ' αυτού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Τζον. Επόμενος αγορητής θα ήταν ε, η καθηγήτρια Βέριτσα Τρίστεντζακ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχε όμω κατεπίγουσε συνεδριάσεις, ανηλυμένε υποχρέωσει, δεν μπόρεσε να φύγει από το Λουξεμβούργο. Θα περάσουμε στου δύο επόμενου ε, αγορητέ ε, και για τον κανονισμό Ρώμη 1 σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών Αγοραπολισιών θα ήθελα να σας πω αν κάποιος θέλει να παρέμβει να συμπληρώσει το δελτίο ε, υποψήφιων αγοριτών ώστε να γνωρίζουμε πόσοι θα θέλουν να παρέμβουν κατά το τέλος της συνδιάσκεψης. Ε, στρέφομαι στον κύριο Hans Schultenberg και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Osnabrück. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας. Έργο μου είναι επ' αυτού να προσπαθήσω να επεξηγήσω τα της προστασίας των καταναλωτών υπό αυτό το εμπορικό δίκαιο. Και όπως είπε ο Σερ Τζον Τόμας πάρα πολύ σωστά, θα πρέπει να συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά με το εφιστάμενο σύστημα το οποίο ισχύει στα κράτη-μέλη. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι έχετε ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο θέλει να πουλήσει σε όλους τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο είναι το δίκαιο το οποίο θα πρέπει να ισχύει για τις συμβάσεις αυτές πώλησης. Τέσσερις είναι οι δυνατότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές. Ενδεχομένως να έχουμε το δίκαιο του καταναλωτή, το δίκαιο του πολιτή ή το συνδυασμό των δύο αυτών δικαίων. Ουσιαστικά μοιάζει κάπως με λοταρία, είναι κάπως τυχαία η επιλογή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει κυρίως με το αν η δραστηριότητα αυτή, η συναλλαγή, στρέφεται προς τον καταναλωτή στη χώρα την οποία είναι κατεστημένος ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται η πιο πιθανή έκβαση θα είναι αυτή που βλέπετε στην τρίτη σειρά της διαφάνειας, δηλαδή ο συνδυασμός των δύο δικαίων, δίκαιο του καταναλωτή, δίκαιο του εμπόρου. Δηλαδή, ο έμπορος μπορεί να επιβάλλει το δικό του το δίκαιο, αλλά παράλληλα ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει διατάξεις του δικού του δικαίου που τον προστατεύουν καλύτερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη για όλους τους εμπλεκομένους. Αν λοιπόν οι επιχειρήσεις θέλουν πραγματικά να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά, αν χρησιμοποιήσουν το εφιστάμενο σύστημα, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αποκεντρωμένο σύστημα το οποίο ήδη ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην περίπτωση αυτή θα ισχύει μόνο το δίκαιο του καταναλωτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο κεντρική στρατηγική, όπου έχουμε δύο επιλογές εδώ, να μην επιλεχθεί δηλαδή κανένα δίκαιο, θα επιβάλλεται πάντα δηλαδή το δίκαιο του καταναλωτή με συγκεκριμένε εξαιρέσει ή σε άλλη περίπτωση αν ο πολιτής θέλει να επιβάλλει το δικό του το δίκαιο, τότε προβλέπεται η εφαρμογή δύο δικαίων, η συνδυασμένη εφαρμογή δύο δικαίων. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, μπορούμε να έχουμε και μία τρίτη επιλογή, μία τρίτη εναλλακτική. Παράλληλα δηλαδή με τις δύο αυτές παραδοσιακές εναλλακτικέ. Δηλαδή, μία μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων σε συνδυασμό με το δίκαιο του εμπόρου που ισχύει σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Στην πράξη αυτή, τα πράγματα θα είναι βέβαια πολύ πιο εύκολα για τον πολιτή. Θα πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίζεται αν θα ακολουθηθούν οι διατάξεις του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων ή οι διατάξεις του δικαίου του πολιτή. Α δούμε τώρα ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά τη κάθε κατάσταση. Α πάρουμε καταρχά το εφιστάμενο καθεστώ, δηλαδή το εναλλακτικό σε σχέση με το μελλοντικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων, όπου επικεντρωνόμαστε στο δίκαιο των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή, αν ακολουθήσουμε το καθεστώ τη Ρώμη 1, ο καταναλωτή είναι σίγουρο ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προστατευτικέ διατάξει στα πλαίσια του εθνικού δικαίου και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χάσει την προστευτική αυτή, τις προστευτικές αυτές διατάξεις προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι καταναλωτές καλύπτονται μόνο από το δίκαιο του πολιτή αν προχωρήσουν σε εμπορικές συναλλαγές διασυνοριακά στο εξωτερικό. Ενδεχομένως βέβαια ο καταναλωτής να πάει στο εξωτερικό για να κάνει εκεί πέρα κάποιε συναλλαγέ, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο προστασία θα είναι το ίδιο με το επίπεδο προστασία το οποίο έχει στη χώρα του. Ακόμα και αν το επίπεδο προστασία τη άλλη χώρα είναι υψηλότερο. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή στην περίπτωση αυτή αν θα μπορεί να εφαρμοστεί το δίκαιο τη αλλοδαπή. Ο καταναλωτή θα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύεται από το Εθνικό Δίκαιο Προστασία του Καταναλωτή. Τώρα, ας δούμε τα θετικά και τα αρνητικά για τους ε, πολιτές. Οι πολιτές ε, οι οποίοι θέλουν ε, να προχωρήσουν στις συναλλαγές με καταναλωτές σε άλλες χώρες που υπάρχει μια χαμηλότερη προστασία, δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν μια καλύτερη προστασία, υψηλότερη δηλαδή από αυτή που προβλέπεται από τη δική τους νομοθεσία και πολύ συχνά οι πολιτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εθνικά συστήματα προστασίας των πολιτών, των καταναλωτών με συγχωρείτε, τα οποία δεν γνωρίζουν και τα οποία διαφέρουν πάρα πολύ από τα δικά τους εθνικά συστήματα. Αυτό προκαλεί βέβαια ένα πρόβλημα για την ε, αρμονική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων η κατάσταση αυτή βελτιώνεται. Ακούσαμε και τα όσα είπε σχετικά ο Σέρ Τζον Τόμας η βασική ιδέα στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων και το βλέπουμε αυτό και στην πρώτη εκδοχή τη πρόταση, ο καταναλωτή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χαίρει ενό υψηλού επίπεδου προστασία. Το υψηλό επίπεδο προστασία θα κατοχυρώνεται σε όλε τι χώρε και δεν θα είναι ούτε αυθαίρετο ούτε τυχαίο. Θα το εγγυάται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει προφανώς το επίπεδο αυτό προστασίας να είναι υψηλότερο από το εφιστάμενο καθεστώς προστασίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, οι καταναλωτές οι οποίοι δεν εμπιστεύονται το δικό τους εθνικό σύστημα θα έχουν αν μη τι άλλο τώρα τη διασφάλιση ότι μπορούν να προστατευθούν από ένα πανευρωπαϊκό σύστημα υψηλότερης προστασίας του καταναλωτή. Βέβαια υπάρχει και ένα μειονέκτημα στο σύστημα αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεκριμένες διατάξεις ε, του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων μπορεί να είναι λιγότερο προστατευτικές για τον καταναλωτή από ότι κάποια εθνικά μέτρα, από ότι κάποιες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσουμε τα σημεία αυτά λίγο αργότερα στη σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχουν πάντως τα σημεία αυτά τα οποία δημιουργούν μια κάποια αβεβαιότητα, τουλάχιστον για την πρώτη μεταβατική περίοδο. Για τους πολιτές η κατάσταση θα είναι καλύτερη, γιατί ε, οι πολιτές θα είναι σε θέση, οι έμποροι θα είναι σε θέση να οργανώσουν ομοιόμορφα πλέον ε, τις συναλλαγές τους, δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να προσαρμόζονται σε διαφορετικά εθνικά συστήματα, καθότι θα υπάρχει ενιαίο σύστημα προστασίας του καταναλωτή και αυτό με τη σειρά του θα προωθεί περισσότερο και την εμπορική δραστηριότητα των ε, πολιτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει επίσης σε μείωση του κόστου, σε μείωση των δαπανών Θα πρέπει πάντως ε, τα πράγματα να είναι κάπως πιο σαφή. Όσον αφορά δηλαδή τους πολιτές εκείνους οι οποίοι προσφέρουν ποιοτικά αγαθά και ποιοτικέ υπηρεσίες και ουσιαστικά δεν φοβούνται τις ε, προστατευτικές για το καταναλωτή διατάξεις. Υπάρχουν βέβαια άλλοι πολιτές οι οποίοι θα προτιμούσαν να διατηρήσουν το εθνικό σύστημα, το εφιστάμενο σύστημα και οι οποίοι θα πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίσουν βέβαια πολλά διαφορετικά εθνικά συστήματα προστασίας του καταναλωτή. Πάντως μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων θα προωθήσει τις πιο ανταγωνιστικές και ποιοτικέ επιχειρήσεις. Προβλέπεται επίσης στο σύστημα αυτό μια πολύ μεγαλύτερη περίοδος υπαναχώρησης και αποζημίωση του καταναλωτή από ό,τι προβλέπεται στα εφιστάμενα εθνικά συστήματα. Σίγουρα υπάρχουν επιμέρους σημεία στην πρόταση που θα πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου η πρόταση αυτή να αποτελέσει μια σωστά λειτουργούσα νέα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία αυτά που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη δικιά μου τη μελέτη, αλλά και σε άλλες μελέτες, έχουν δοθεί πολλά παραδείγματα. Όπως είπε και ο Σερ Τζον Τόμας, υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία στην υφιστάμενη πρόταση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων, τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη δυνατότητα opt-out η οποία προβλέπεται. Αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε όμως το κείμενο αυτό, τότε πιστεύω ότι πραγματικά θα καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ καλή νομοθεσία. Θα έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων που θα αποτελέσει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία υπέρ των καταναλωτών και θα κάνει τελικά την ε, ποιοτική, μάλλον θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο ορατή και πολύ πιο ποιοτική ουσιαστικά στα μάτια των καταναλωτών και των εμπόρων. Σας ευχαριστώ. Μαρτίν Μπεάτισε, κυρία καθηγήτρια, είτε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να καταφέρει κανείς ε, αυτό το δίκαιο των συναλλαγών να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει σε σχέση με τις, ε, σε με τις διατάξεις Ρώμης 1 να είναι σαφής. Αυτό το δίκαιο θα μπορούσε να καθοριστεί είτε ένα ενιαίο δεύτερο καθεστώς σε σχέση με το δίκαιο. Ο καθορισμός ως ένα δεύτερο καθεστώς ε, εγχώριου δικαίου θα μπορούσε να οδηγήσει στο να εφαρμοστεί χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα αυτών των διατάξεων διασυνοριακά σε συναλλαγές. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την νομιμότητα αυτού του ισχυρισμού κάποιοι συγγραφείς αρνούνται την ικανότητα να απορρέει εθνικό δίκαιο από αυτό το δυναμικό. Άλλοι διαρωτώνται για τις επιπτώσεις που ενώ θα καθορίζεται ως εγχώριο δίκαιο με ε, επιτόπιες ερμηνείες θα μπορούσαν εδώ να αφορώνται μελλοντικές οδηγίες. Όλα, αυτά τα σκεπτικά και σκέψεις δίνουν το μέσα να αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχει ένα υβρίδιο εδώ, είναι υβριδιακή η φύση αυτού του δικαίου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ του κελίφους και του περιεχομένου. Το κέλυφος πρέπει οπωσδήποτε να συνδράμει την δευτερογενή ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό υπό τον όρο Ευρωπαϊκής Ερμηνείας και υπό τον έλεγχο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 10. Το περιεχόμενο τώρα σε σχέση με την ρύθμιση των συναλλαγών είναι ένα δεύτερο σκέλος και δικαιώνει για παράδειγμα σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών που πρέπει να διασφαλίζεται σε ίσο επίπεδο με την προστασία εκείνη που παρέχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Τώρα, σε σχέση με το, τις ρυθμίσεις Ρώμης 1 ε, συνάγεται από το δευτερογενές αυτό καθεστώς ότι οι διατάξεις Ρώμης 1 θα μπορούν να ε, εφαρμόζονται και να ισχύουν ομαλά και κανονικά. Δεν επιλέγει κανείς ε, ε, με το όργανο αυτό υπάρχουν δύο φάσεις. Αφενός υπάρχει επιλογή όσον αφορά νομοθεσία κράτους μέλους και του ενισχύ δικαίου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει επιλογή του ευρωπαϊκού δικαίου συναλλαγών υπό το εθνικό πλαίσιο. Μπορεί κανείς να επιλέγει το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο ε, χωρίς να υπάρχει ρητή ε, διάταξη γι' αυτό. Όμως αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει βούληση επιλογής αυτού του δικαίου από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του με το δίκαιο αυτό δεν θα υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ των διατάξεων που θα αφορούν την νομοθεσία κρατών μελών σε αυτό το πεδίο. Το άρθρο 6.2 των διατάξεων της Ρώμης ε, που προβλέπει διαφορετικό επίπεδο προστασίας καταναλωτών ε, δεν θα έχει εδώ πρακτική σημασία. Υπάρχει εξουδετέρωση θα έλεγα σε σχέση με τις διατάξεις αυτές όσον αφορά το εθνικό καθεστώς. Ωστόσο όμως μπορεί να εκφράσει κανείς τη θλίψη του για το ότι ένα τόσο σημαντικό σημείο αναφέρεται στα σκεπτικά ή στις αιτιολογικές σκέψεις σε σχέση με τον κανονισμό και το επεξηγηματικό υπόμνημα. Καλύτερο θα ήταν να είχε ενταχθεί στα άρθρα, σε άρθρο του κανονισμού αν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο άρθρο 11. Στο άρθρο 11 περί τίνος πρόκειται θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο κείμενο, στη διατύπωση, τους όρους που βρίσκονται με κόκκινο στο κείμενο, για να είναι σαφέστερες οι διατάξεις σε σχέση με το ευρωπαϊκό αυτό δίκαιο για συναλλαγές. Σε σχέση με τις άλλες ε, υποχρεωτικές ε, προβλέψεις ε, αφορούν το πρώτο καθεστώς που εντάσσονται στο ίδιο εύρος των διατάξεων του δευτέρου καθεστώτος του CESL. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ε, δέσμευση όσον αφορά το, το αιτιολογικό 27, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό ανισοτήτων από το εύρος εφαρμογής του CESL. Αυτός ο αποκλεισμός, αυτή η εξαίρεση αφορά ήδη τις διατάξεις ε, που προβλέπουν την ε, ε, συμμετοχή σε, αυτή, σε αυτό το σκέλος. Στο γαλλικό δίκαιο για παράδειγμα, οτιδήποτε αντιβαίνει τις υποχρεωτικές διατάξεις θεωρείται παράνομο. Ο κίνδυνος ποιος είναι, ότι θα μπορεί να αποκλείεται κάτι από το εύρος του ΣΕΣΛ και να εφαρμόζεται και να, σε σχέση με την επιλογή των ε, ε, μερών να ε, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η ανισότητα θα πρέπει να, είναι, να περιορίζεται ώστε να μην οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αυτός ο μηχανισμός ο οποίος θα θεσπίζεται θα πρέπει να εγκρίνεται από τη στιγμή εκείνη που θα προστατεύεται από τους υποχρεωτικούς δεσμευτικούς ε, κανόνες και κανονισμούς του δεύτερου καθεστώτος ε, υψηλού βαθμού, υψηλότατου ε, επίπεδου προστασίας. Στο ενημερωτικό έγγραφο μπορείτε να δείτε συγκριτικούς πίνακες που συγκρίνουν την εθνική νομοθεσία και εθνικές διατάξεις σε σχέση με το τι ισχύει με το ΣΕΣΛ θα δείτε πολλές φορές ότι παρέχεται περισσότερη προστασία από το ΣΕΣΡ έναντι του εθνικού δικαίου. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων ήρθατε ε, ζητώ συγγνώμη που δεν το προανέφερα Στη συνέχεια για την προπαρασκευή των συνοδευτικών μέτρων όσον αφορά τέτοιου είδου συμβάσεις από τον κύριο καθηγητή Dirk Staudenmayer, επικεφαλής της διεύθυνση για την Δικαιοσύνη για το Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθηγητά, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ε, το σχέδιο για το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων εξέδωσε και μία ανακοίνωση που εξηγεί το πολιτικό πλαίσιο και τους στόχους της πρότασης, αλλά και έναν αριθμό συνοδευτικών μέτρων. Ο στόχος αυτών των μέτρων ήταν να γίνει πιο εύχρηστη και πιο χρήσιμη στην πράξη αυτή η πρόταση. Και αναφέρονται διάφορα τέτοια συνοδευτικά μέτρα. Όλος ιδιαίτερος αναφέρεστε και εσείς στο ευρωπαϊκό μοντέλο συμβατικών όρων. Και η Νταϊάννα Γόλης είναι εδώ φυσικά και ε, σας θυμίζω ότι κατόπιν δική στις πρωτοβουλίες ε, συμπεριλήφθη αυτό το σημείο στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την σχετική πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, λοιπόν, περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο. Ένας πολίτης μπορεί να πωλήσει τα αγαθά του στις υπόλοιπες 26 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο δίκαιο, μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτός είναι ο στόχος, ε, δηλαδή ε, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο συμβατικών όρων. Στο ιδανικό, στην ιδανική περίπτωση ε, ε, προσθέτεται μόνο τα ονόματα των συναλλασσομένων, ε, το, τις ποσότητες των αγαθών, την τιμή και την ημερομηνία ίσως παράδοσης. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο γιατί τα υπόλοιπα θα είναι ρυθμισμένα. Ο στόχος λοιπόν αυτού, το, αυτού του ευρωπαϊκού μοντέλου συμβατικών όρων ουσιαστικά είναι να ε, δίνουμε μόνο τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένη ε, συναλλαγή, αλλά να ισχύουν ούτως ή άλλως κάποιοι όροι ε, για τα συναλλασσόμενα μέρη. Παραδείγματο χάρη σε από επιχείρηση σε επιχείρηση. Βλέπω εδώ μια σύμβαση που προβλέπει ότι θα πρέπει να εξακριβωθεί η ποιότητα των αγαθών και θα πρέπει να γίνει η εξέταση αυτή σε μια εύλογη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Ε, αυτό για την επίτευξη της νομικής ε, ασφάλειας ως έσχατο μέσο για την εξασφάλιση αυτής. Βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να προσδιορίσουν ε, τη διάρκεια αυτής της περίοδου επακριβέστερα. Παραδείγματος χάρη να αποφασίσουν θα είναι δύο, τρεις, τέσσερις ημέρες σε συνάρτηση με τις ανάγκες τις δικές τους του κλάδου και της φύσης των προϊόντων. Είναι το αντικείμενο της συναλλαγής. Δηλαδή, οι κανόνες ε, της δικής μας πρότασης, βλέπουμε σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα πώς θα μεταφέρονταν σε μία σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα συντάξει αυτό το σετ κανόν μόνη τη, αλλά σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους. Εκείνοι πρέπει να καταθέσουν προτάσεις γιατί εκείνοι θα χρησιμοποιήσουν τους κανόνες. Εμείς διευκολύνουμε μόνο την διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο το πρώτο συνοδευτικό μέτρο. Το δεύτερο αναφέρθηκε και αυτό ε, προηγουμένως ε, για το άρθρο 14 του βασικού κανονισμού. Ε, συγκρότηση βάσης δεδομένων συγκεκριμένα. Μια βάση δεδομένων όπου όλα τα κράτη-μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελεσίδικες αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων τους που εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό Σέτη κανονών διότι είναι άμεσα εφαρμόσιμο ενωσιακό δίκαιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο δικαστής ε, στο Τούρκο ή στην ε, Νάπολη ε, δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί να πει ένας δικαστής ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, για αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη ε, πρέπει να αποφασιστεί κάτι από τους συναδέλφους μου σε κάποια άλλη χώρα. Μπορεί να συμβουλευτούν λοιπόν τη βάση δεδομένων και θα υπάρχουν επιγραμμικά και μεταφρασμένες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Άρα μπορεί να κάποιος που είναι στο Τούρκο να βρει την απόφαση του συναδέλφου του δικαστήριου Στη στην πολύ σε μία ε, παρεμφερή υπόθεση και μπορεί να αποφασίσει ο δικαστής ειδού Θα αποφασίσω και εγώ το ίδιο αν κρίνω ότι είναι λογική η δική του απόφαση. Αυτό που θέλουμε είναι μία de facto σύγκληση της ερπινίας των αθηνικών δικαστηρίων στο μέτρο που πρόκειται για ε, άμεσα εφαρμόσιμο δίκαιο. Αυτή η βάση δεδομένων δεν θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα δικαστηρία, αλλά για όλα τα συμβαλώμενα ενα μέρη για το κοινό όλοι όσοι θα εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και για λόγους πλήρους διαφάνειας να έχουν πρόσβαση στην πλήρη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων που ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το ενιαίο σετ κανόνων. Αυτό είναι το δεύτερο μέτρο. Τρίτο συνοδευτικό μέτρο, επίσης το έχετε ήδη αναφέρει, είναι κοινή κανόνες. Ζητήσαμε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων να προετοιμάσουν την μελέτη αντικτύπου αλλά και την σύνταξη κοινών κανόνων στο άμεσο μέλλον ο στόχος είναι να επικουρήσουμε τους συνομοθέτες ε, στην ε, νομοτεχνική διαδικασία αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τους χρήστες, τα συμβαλόμενα μέρη δηλαδή που θα κληθούν να εφαρμόσουν ε, τους κανόνες του νέου ευρωπαϊκού δικαίου. Κατάρθρο θα προσφέρουμε επεξήγηση ερμηνεία της προθέσεως του νομοθέτη. Για ποιο λόγο συμπεριέλαβε στο νομοθέτημα αυτή τη διάταξη και θα δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε στην πράξη πώς λειτουργούν αυτές οι διατάξεις με τρόπο ώστε τα συμβαλόμενα μέρη να έχουν και ε, το δίκαιο στη διάθεσή τους αλλά και κάποιες ε, διευκρινήσεις ε, για τον δίκαιο τόσο ώστε να είναι πιο εύχριστο στην πράξη. Τέταρτο συνοδευτικό μέτρο, που, κάτι που έχει ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μήνα μετά την έκδοση της αρχικής απόφασης. Ε, μία πρόταση λοιπόν για μία οδηγία για την ε, εναλλακτική επίλυση διαφόρων ε, και για την επιγραμμική εναλλακτική επίλυση διαφορών. Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Αυτές οι δύο προτάσεις εξεδόθησαν μία, ένα μήνα μετά την αρχική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ο στόχος είναι να ρυθμίζουν ένα πρόβλημα που επίσης έχουν εντοπίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή δυσκολία σε σχέση με την ε, ε, πανόρθωση ζημιών σε διασυνοριακό επίπεδο, σε διασυνοριακές συναλλαγές ε, και προχωρήσαμε πολύ γρήγορα ευτυχώς διότι αναγνωρίσαμε ότι πρόκειται για δύο προτεραιότητες για μας Εάν εφαρμοστούν σωστά αυτές οι προτάσεις, ε, ε, τα συμβαλόμενα μέρη σε κατάσταση διασυνοριακής διαφοράς θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να προσφύγουν στα δικαστηρία σε ε, συναλλαγή από επιχείρηση σε ιδιότητα, αλλά και να προσφύγουν σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών στον εναλλακτικό στο εναλλακτικό σύστημα επίλυση διαφορών. Επόμενο συνοδευτικό μέτρο που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μα είναι η υποστήριξη τη κατάρτιση. Ο καθηγητή Μπερλίνγκουερ που είναι ένα από του συζητητέ του κοινού ευρωπαϊκού ε, δικαίου πολίσεων, ε, ήταν ένα από αυτού που μα ενέπνευσε την ιδέα αυτή, δηλαδή να ε, προσφέρουμε κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά όχι μόνο και των καταναλωτών και των ε, επιχειρήσεων για να προωθήσουμε αυτή την πρόταση. Δηλαδή το ευρωπαϊκό δίκαιο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο, ξαναλέω, κατάρτισης για τους επαγγελματίες αυτού του τομέα, ε, ούτως ώστε να δίνονται προσφορότερες συμβουλές. Όλα αυτά τα συνοδευτικά μέτρα υπάρχουν ήδη και ο στόχος ε, δεν είναι να έχουμε μόνο και μόνο ένα ενιαίο δίκαιο βάση του οποίου μπορεί να εξάγει η επιχείρηση τα αγαθά της, αλλά αυτό το ενιαίο δίκαιο να μπορεί με ιδιαίτερη ευκολία να χρησιμοποιείται στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι καθηγητά Στάουντεν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσει και οι παρουσιάσεις, η τροφή για σκέψη και από πλευράς του, 10, ε, από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέως ε, έχει αφήσει ε, λόγω της απουσίασης έχει αφήσει το έντυπο με τον λόγο που θα εκφωνούσε. Έχουμε τώρα ευκαιρία τα μέλη της Επιτροπής και των Εθνικών Κοινοβουλίων να διατυπώσουν ερωτήσεις ή να κάνουν σχόλια στις παρεμβάσεις τους. Έλαβα μόνο ένα αίτημα να παρέμβει κάποιος μέχρι τώρα. Υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ε, θα ήταν καλό απλά να αναφέρατε την επιθυμία σας ε, να παρέμβετε. Αλλά μόνο και μία γραπτή, ένα γραπτό αίτημα υπάρχει. Να μην πιστεύει κανείς ότι υπάρχει εθνική προτίμηση δίνοντας τον λόγο στον, στον κύριο Άλαν Μπίφ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι θέμα εθνικής προτίμησης. Πρόεδρε, έχοντας ακούσει μια τέτοια εξαιρετική ομάδα παρεμβάσεων στις εισηγήσεις, ίσως θα είναι καλά μαντάτα ότι από τα εθνικά κοινοβούλια πολλοί από εμά ε, δεν ανοιχνεύσαμε ακόμα το επίπεδο ενθουσιασμού που ένα τέτοιο εγχείρημα θα προκαλούσε, που ένα τέτοιο εγχείρημα με τέτοια προτερήματα θα μπορούσε να εγείρει. Και από πλευρά ε, της Βρετανικής ε, ανταπόκρισης υπήρχε μάλλον μια πιο τριοπαθήσα ε, ή ας το πω έτσι μεγαλύτερων επικρίσεων άρνηση προς αυτό το εγχείρημα. Για τη διευκόλυνση τώρα για την ενιαία εσωτερική αγορά και τη διευκόλυνση για τον, το πλαίσιο των ε, συναλλαγών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις πολλά βάρη υπάρχουν, ε, πολλές φορές βάρος φορολογικό ή άλλου είδους. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια εναλλακτική δυνατότητα σε όλες αυτές τις δυνατότητες τότε συναλλαγών. Όμως εξεπλάγει όταν είδα τις ε, αντιδράσεις σε σχέση με αυτό το εγχείρημα στο πλαίσιο όπου ε, οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, ε, νομικοί φορείς και όργανα, μια τέτοια δαπανηρή διαδικασία είναι αυτή που δεν θα ήθελαν, δεν θα επέλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν και φυσικά δεν είναι μόνο θέμα επιλογής καταναλωτών αλλά και το θέμα επιλογής επιχειρήσεων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί και θα ήθελα απλά και μόνο να αναφέρω ως επιφύλαξη αυτό τον όρο, αυτή την προϋπόθεση. Και από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Ίσως δεν αναφέρεται τόσο, τόσο συχνά η ανάγκη εναρμονισμού του εθνικού δικαίου σε αυτό το πλαίσιο. Εναρμονισμού και προσαρμογής, αντί να υπάρξει ένα πρόσθετο μέσο το οποίο δεν θα χρησιμοποιούν συχνά οι πολίτες. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ποιος άλλο θα ήθελε να παρέμβει, παρακαλώ. Κάνοντας αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να μας αναφέρετε το όνομά σας, την χώρα προέλευσή σας και τη Βουλή που εκπροσωπείτε. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορώ το, τα μηνύματα νοηματικά να τα κατανοήσω από εδώ. Δεν βλέπω να επιθυμεί κανείς να παρέμβει. Όλοι νομίζω έχουμε συντριπτικά πιστεί από τις παρεμβάσεις που έγιναν. Και αν επιτρέπετε, εγώ θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ τώρα. Και έχουμε να ακούσουμε πρώτα τους ε, οι ε, του πάνελ αυτού και μετά να έχουμε μια γενικότερη συζήτηση, ευρύτερη συζήτηση. Ίσως αυτό θα έδινε την ευκαιρία, έχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης, να συμπεριλάβουμε και διάφορες άλλες πτυχές από ε, αυτόν. Πρόεδρε, εσείς είστε ο πρόεδρος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Είναι εξαιρετική ιδέα θα έλεγα αυτή και για την ε, σύνοψη των ε, παρεμβάσεων ε, δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα μπορούσα εγώ να συνοψίσω τα, τις παρατηρήσεις των εξεχόντων ε, αγοριτών. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον καθηγητή Ζένσμπουργκ, Πάτρικ Ζένσμπουργκ, ε, από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, εκείνο να αναλάβει την Προεδρία ω συντονιστή αυτού του δεύτερου πάνελ. Σα ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση, που πραγματικά το εκτιμούμε ιδιαίτερα και είναι πολύ αξιόλογη. Σα ευχαριστώ πολύ που ε, λαμβάνετε την προ... λάβατε την Προεδρία ε, ως ε, συντονιστής του πρώτου πάνελ. Παρακαλώ καθηγητά Σένσμπουργκ να λάβετε εσείς τώρα τον λόγο και να προεδρεύσετε εσείς ως συντονιστής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω, αν επιτρέπετε, για το ότι τόσο γοργά δίνετε τον λόγο στο δεύτερο πάνε, στο δεύτερο γύρο. Υποθέτω ότι αναμένουν τα ερωτήματα κάπως περισσότερο να απαντηθούν. Δεν είναι αυτό επαρκές ακόμα σήμα, δεν σηματοδοτεί επαρκή συνένεση. Είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ε, και απόψεων που απαιτείται και ίσως μετά το δεύτερο αυτό πάνε, το δεύτερο γύρο, να ξεκινήσουμε συζήτηση, γενικότερη συζήτηση. Διότι το δεύτερο πάνελ υπόσχεται ότι θα γύρει το ενδιαφέρον στον τρόπο προσέγγισης και νομικά υπονομική πτυχή αλλά και των εφαρμογών στην πρακτική εφαρμογή και έτσι με αυτή την επιλογή θα πρέπει με αυτό να δούμε ότι από πλευρά τη ε, Γερμανική ε, Ομοσπονδική Βουλή ε, δεν είναι μόνο το θέμα τη επικουρικότητα. Χαιρόμαστε για το έργο τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και για το έργο τη Επιτροπή επαυτών. Ελπίζουμε ότι με αυτό το έναυσμα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη θετική πορεία. Συγχαίρουμε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με τον, για τον έντονο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και είμαστε ευγνώμονε για το γεγονό ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε και να ενταχθούμε σε αυτό το πλαίσιο και εμεί απόψε εδώ. Ο πρώτο που θα παρέμβει ο καθηγητή καθηγητή Στέφαν Φόγενάουερ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Του δίνω τον λόγο για να κάνει την παρουσίασή του, παρακαλώ. Κύριε Φόγενάουερ, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω σε σχέση με την σύνταξη και διατύπωση αυτού του δικαίου το στυλ ρενταξιονέλ όπως θα έλεγαν οι Γάλλοι, ε, δηλαδή διατυπωτικό ύφος ε, ή τις νομικές διατυπώσεις επί των διατάξεων ώστε να μπορέσουν να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Εδώ υπάρχουν και τα θέματα της δυσχέρειας ε, μετάφρασης, με, δια, ικανοποιητικής μετάφρασης όλων αυτών των έννοιων. Και θα αναφέρω κάποια στοιχεία όσον αφορά τις, ε, τα παραδείγματα θα βρείτε αρκετές δυνατότητες στο σημείωμα και σε σχέση με αυτά τα οποία προηγούμενα ο Σετζόν ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής σας. Εισαγωγικά τώρα απλά θα ήθελα να πω τούτο. Όλοι γνωρίζουμε το προαιρετικό αυτό μέσο το οποίο ε, ως σημείο κίνησης διαφέρει από το συμβατικό πλαίσιο ε, το εθνικό της νομοθεσίας και θα πρέπει να θέλει να είναι ελκυστικό για τους χρήστες να επιλέξουν οι χρήστες να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Λαμβάνοντας αυτή την απόφαση θα επηρεαστούν σίγουρα από την ποιότητα διατύπωσης ε, των διατάξεων οι συμβαλόμενοι. Αυτό μπορεί να είναι θελκτικό ή και να είναι και αποτρεπτικό θρεπτικό σε σχέση με του χρήστε. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά πρέπει να είναι καλύτερο το επίπεδο αυτό από τα υφιστάμενα πρότυπα, ώστε να έχουν προτίμηση να το επιλέξουν οι συμβαλόμενοι. Διότι όπως γνωρίζουμε από, για τις επιλογές όσον αφορά το δίκαιο στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική ζωή, δεν είναι, ε, είναι η εξοικείωση με το μέσο και η ποιότητα. Και για να ξεπεράσουμε την ε, αδράνεια που κάνει τους ε, χρήστες να επιλέγουν εκείνο το οποίο γνωρίζουν καλύτερα, πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη διατύπωση και στην αποσαφήνιση πραγμάτων. Και αν όλα αυτά δείχνουν κάπως ανίκια ή αισθάνονται οι χρήστες ότι είναι ανίκια για αυτούς, τότε θα παραμείνουν στα εθνικά πλαίσια δικαίου και δεν θα ε, προσελκυστούν από αυτό το νέο μέσο. Λοιπόν, σε σχέση με τους γενικούς όρους ε, αναγνωρίζεται αυτό από την Επιτροπή και συχνά γίνεται λόγος να υπάρχει ένα φιλικό προς τους χρήστες μέσο. Η φιλικότητα προς τους χρήστες λοιπόν είναι ο πύχης, είναι ο γνώμονας. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει, καθώς γνωρίζουμε από την Επιτροπή, απλή και εύληπτη γλώσσα. Σημαίνει ένα μέσο το οποίο θα είναι σε θέση να κατανοήσουν εξίσου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές χωρίς την πραγματογνωμοσύνη ενός νομομαθούς ε, συμβούλου ή ενός ε, δικηγόρου. Τώρα, σε σχέση με την επικέντρωση για τις προτάσεις για βελτίωση, διότι δεν είναι έργο μου να επενέσω αυτό το οποίο επετέφθη, αλλά να προτείνω επικοδομητικά κάποιες ε, επικρίσεις ή προτάσεις ε, ε, κριτικού χαρακτήρα. Σε σχέση λοιπόν με αυτό θα ήθελα για τα πρακτικά να πω ότι δεν συμμερίζομαι επί παντός όλες τις απόψεις, αλλά έχω με ιδιαίτερο θαυμασμό και εκτίμηση για τους, την ικανότητα των νομομαθών που έχουν συνεισφέρει, αλλά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και διατυπωτικά θα αναφερθώ σε αυτές. Όσον αφορά ε, ε κάποιους που ενδιαφέρονται σε σχέση με ταινίε του Hollywood, θα ε, κατανείμω τις παρεμβάσεις μου μεταξύ των καλών, των κακών και των άσχημων. Ξεκινώντας με τους καλούς, το θετικό πρόσημο και το κυριότερο θετικό της πρότασης είναι η εύληπτη και προσπελάσιμη γνώση, γλώσσα, με συγχωρείτε. Βρίσκεται σε ένα εύθετο επίπεδο στοιχείων. Δεν είναι ούτε υπερβολικά σχολαστική, ούτε γενική ή αφε, ε, γενικόλογη όσον αφορά τα στοιχεία. Αυτό δίνει ένα θετικό συμβιβασμό μεταξύ των παραδοσιακών διατυπωτικών προτύπων που έχουμε στα εθνικά μας συστήματα νομοθεσίας στην Ευρώπη, που θα πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης και της νησιωτικής Βρετανίας. Ένα άλλο θετικό στοιχείο, αλλά αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο και υπάρχουν παγίδες εδώ, είναι ότι παγίδα, το κείμενο αφήνει πολύ περιθώριο για ερμηνεία ή ερμηνευτικό περιθώριο ή δυνατότητες προσαρμογής ως προς κάποια πρότυπα. Τώρα, υπό αυτούς τους όρους Όσον αφορά τα αρνητικά υπάρχουν κάποια δομικά διαθωτικά προβλήματα τα οποία απορρέουν λόγω αποφάσεων, πολιτικών αποφάσεων όσον αφορά την διατυπωτική ε, προσέγγιση από πλευράς ε, ε, γλώσσας που δεν έχει σχέση με τα θέματα ουσίας. Η χρήση συχνά αφηρημένων ή γενικόλογων όρων θα πρέπει να παραμένει σε ένα περιορισμένο πλαίσιο. Το άρθρο 3 προβλέπει την υποχρέωση των συμβαλωμένων να συνεισφέρουν στον στόχο που αναμένεται, στην επίτευξη του αναμενόμενου στόχου. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικόλογο όσον αφορά αυτό το αμφίσιμο καθήκον και ίσως αρχικά προτού υπάρξει η νομολογία η οποία θα είναι ε, προσβατή στους ε, δικαστές ε, και στην Νεάπολη της Ιταλίας αλλά και στο Τάκου της Φινλανδίας θα υπάρχει σημαντική νομική αβεβαιότητα. Δεν θα γνωρίζουν υποχρεωτικά οι εμπλεκόμενοι οι συμβαλόμενοι που θα βρίσκονται. Προφανώς αυτά τα προβλήματα συνδέονται με την παρατήρηση που έγινε προηγούμενα. Αν θέλουμε να έχουμε υψηλό βαθμό ελαστικότητας είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε βαθμό νομικής βεβαιότητας και ασφάλεια. Τώρα, σε σχέση με τα εθνικά συστήματα πρέπει να δούμε ότι δυσχεραίνεται αυτό το εγχείρημα μέσα σε ένα πολυγλωσσικό καθεστώς πολυεθνικού πλαισίου όπως στην Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σοβαρό λοιπόν αυτό το πρόβλημα από ότι αν υφίστατο μόνο σε ένα εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ επίσης θα υπάρξει ένα πρόσθετο αρνητικό αντικίνητρο που ίσως θα απέτρεπε τους συμβαλόμενους να το επιλέξουν. Προσελ, προσελκύει μάλλον ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τριβές και όχι να, δεν θα βοηθούσε να αποφύγουμε τριβές ώστε να μην έχουν δουλειά οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις αντιπαραθέσεις. Ένα άλλο σημείο, η, η γενικόλογη και αφηρημένη αυτή διατύπωση παρόλους τους μηχανισμούς ε, επιδιατησίας ε, η, θα, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις ε, αρνητικές. Ένα δεύτερο σημείο είναι η χρήση της νομικής ορολογίας όπως προανέφερα, η Επιτροπή θέλει να υπάρχει ένα φιλικό προς τους χρήστες μέσο, το οποίο θα μπορεί να είναι εύληπτο και να κατανοείται χωρίς τη βοήθεια νομομαθών και νομικών ε, πραγματογνωμόνων. Αυτό αποφεύθηκε σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι συνολικά και παντού. Αν δει κανείς την ε, την διατύπωση anticipating non-performance ε, ή ε, περιπλοκές διατυπωτικές που ε, δεν αποσαφηνίζουν τα πράγματα αμφιβάλλω αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ε, εκλογικής περιφέρειας της κυρίας Νταϊάννα Γουόλης θα βρουν ότι αυτό τους βοηθά να πορευθούν προς τη σωστή οδό. Ωστόσο, τέτοιου είδους ε, αβεβαιότητες θα πρέπει να αρθούν. Το δεύτερο πρόβλημα, και αυτό σε κάποιο βαθμό είναι αναπόφευκτο, είναι η χρήση ορολογίας που με μια πρώτη ματιά φαίνεται οικία στον εθνικό χρήστη ο στόχος της ε, σύνταξης ε, διεθνών τέτοιων ε, μέσων είναι να επιτευχθεί μια ουδέτερη συστημικά ορολογία αλλά για τα αποτελέσματα όσον αφορά την ε, ενιολογία, τη σημασιολογία αυτών των πραγμάτων υπάρχει διαφορετική απόχρωση ε, και χρειά όσον αφορά τους ε, Βρετανούς νομομαθείς ή τους Γερμανούς νομομαθείς. Τέτοιου είδους δάνεια εθνικής ορολογίας καθιστούν δύσκολο το να υπάρξει να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ορολογίας σε αυτό το πολυεθνικό πλαίσιο. Για τα άσχημα σημεία της πρότασης όταν μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κατά την νομοτεχνική διαδικασία υπάρχουν παραδείγματα κακής διατύπωσης και οφείλονται κυρίως στη βιασύνη τη σπουδή με την οποία ε, καταρτίστηκε το τελικό σχέδιο. Υπάρχουν περιτά σημεία, ε, έλλειψη συνοχής ανάμεσα σε διάφορες ε, διατάξεις, διάφορα τμήματα του νομοθετήματος και κυρίως ανάμεσα στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές. Επίσης υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο περιπλοκότητας συνήθως που δεν καθιστά το νομοθέτημα εύχριστο φιλικό προ το χρήστη. Πώ λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα έπρεπε να βελτιώσουμε τα κακά σε εισαγωγικά σημεία στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή να είναι πιο συγκεκριμένη, πιο ενεργή η διατύπωση ε, και να χρησιμοποιούμε μία νομική ορολογία ε, γνωρίζοντα σε ποιον αποτινόμαστε. Είτε θα μιλάμε στου επιχειρηματίε είτε στους δικηγόρους, επαγγελματίε. Πρέπει όμω να είμαστε ξεκάθαροι και να ακολουθούμε μία γραμμή κατά τη σύνταξη του κειμένου. Άρα αυτό απαιτεί τροποποίηση, ε, η θελημένη τροποποίηση της ε, πολιτικής που ακολουθείται για τη σύνταξη του νομοθετήματος. Αντίθετα, για να ξεφορτωθούμε τα άσχημα σε εισαγωγικά σημεία, αυτό είναι απλούστερο. Ε, τα επόμενα σημεία ε, θα, ακού, θα διαπιστώσουμε ποια είναι τα περιτά σημεία, οι ασυνέπειες, οι ανακολουθίες κτλ. Αλλά βέβαια χρειάζεται χρόνος ε, για να απαλληφθούν όλα αυτά. Και κάτι που αναφέρθηκε δει σήμερα και είναι σημαντικό είναι ότι αν θέλετε να καταργήσετε την περιπλοκότητα. Θα πρέπει να κάνετε ένα επίσημο σχόλιο προσθέτοντας έτσι ένα επίπεδο ε, περιπλοκότητας ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τους διεθνούς όρους, ε, για τις διεθνείς ε, συμβάσεις, βλέπουμε ότι είναι επιβοηθητική αυτή η όρη, αλλά δημιουργούν μεγαλύτερη περιπλοκότητα και λειτουργούν ορισμένε φορέ ω ε, κίνητρα ε, και δημιουργούνται νέε διαφορέ. Εγώ πιστεύω ότι ε, θα έπρεπε να αποφύγουμε τι ερμηνείε του δικαίου, τα λεγόμενα commons. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Επίσης, να αναδιατυπωθεί πλήρως η πρόταση επιτάπητος για να γίνει αυτό και ξέρω δεν αρέσει στους πολιτικούς. Θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο σε αυτό, να αφήσουμε χρόνο για τον προβληματισμό και για την κατάλληλη διατύπωση. Αν ποτέ εφαρμοστεί αυτή η νέα νομοθετική πρόταση είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να αποφύγουμε την ελλειπή, την ατελή ε, ε, ε, ποιότητα προς τη διατύπωση. Αξιότιμε καθηγητά Φόγεναουερ, εν μέρη παρουσιάσατε τις επιφυλάξεις που από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων διατυπώνονται και εν μέρη υπό το ενδεδειγμένο πλαίσιο αναφέρονται αυτά το, το, τη σκοπιμότητα να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών για τις αγοραπολισίες. Ως επόμενη αγορήτρια έχουμε την κυρία Χάνε Μελίν από μια σε όλους γνωστούς εταιρεία υποθέτω την eBay που επιτυχώς δραστηριοποιείται στην αγορά. Διαρωτώ με τώρα, αν δούμε την πλευρά των επιχειρήσεων, αγαπητή κυρία Μελίν, τότε ένα 28ο τέτοιο καθεστώς θα χρειάζεται για να είναι κανείς πιο επιτυχής σε σχέση με το eBay ή μήπως ε, με απατάει η εντύπωση αυτή και ίσως ε, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει διαφορετικά. Εξηγήστε μας λοιπόν γιατί μια τόσο επιτυχής εταιρεία η eBay και οι οικονομικοί κύκλοι που έχουν επιτυχία και χωρίς το ευρωπαϊκό δίκαιο επί των συναλλαγών, γιατί εσείς θέλετε να υπάρξει αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο επί των συναλλαγών. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ουσιαστικά δεν παρεμβαίνω τόσο από πλευράς ε, των απόψεων και της θέσης της eBay, αλλά από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την eBay όσον αφορά την, ε, τις δράσεις τους ε, και τη δραστηριότητά τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ομιλώ υπό το πλαίσιο διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών είτε στο ηλεκτρονικό εμπόριο είτε των παραδοσιακών συναλλαγών διότι όλες αυτές ε, όλο και πιο όλο και περισσότερο ε, ε, αλληλεξαρτώνται. Πριν από λίγα χρόνια δεν έκαναμε λόγο για ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά μόνο για ε, εμπόριο παραδοσιακά. Κάνουμε λόγο λοιπόν για μεγάλες, μεγάλη ανάπτυξη. Ποτέ δεν ήταν δυνατό να έχει κανείς τόσες ε, συναλλαγές διασυνοριακά. Κατά 126% αυξήθηκαν αυτές οι συναλλαγές από το 2004 ως το 2010 σε σχέση με τις συναλλαγές της eBay. Τεράστιο ποσοστό αύξησης αυτό και σχεδόν 96-98% αυτών που χρησιμοποιούν την eBay από τη Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο εξάγουν. Εξάγουν. Είναι, αφορά και τους μεγαλύτερους πολιτές και τους μικρότερους. Κατά μέσον όρο πολλούν σε πέντε χώρες κατά μέσο όρο πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξάγουν προς αυτές. Έχουμε τα εργαλεία της τεχνολογίας και το διαδίκτυο που μειώνουν τις δαπάνες για τους καταναλωτές. Κινητά τηλέφωνα, τεχνολογικά μέσα τα οποία διευκολύνουν τις επικοινωνίες, αυξάνουν τη διαφάνεια των πληροφοριών και δίνουν τη δυνατότητα στους συμβαλόμενους να αυξήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Και όλα αυτά, γιατί βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ. Οι όγκοι των διασυνοριακών συναλλαγών όμως παρόλα αυτά παραμένουν χαμηλοί. Τα στοιχεία μας μας δείχνουν ότι είναι κάτω από το 20% συνολικού όγκου συναλλαγών. Τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν πολύ μετριοπαθή αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών. 2008-2009 8,8% μετά ναι, ε, το, μέχρι το 2011 9,6% και αυτό γιατί, σε τι οφείλεται και αυτό διότι ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να διασυνδέονται διασυνοριακά οι συμβαλόμενοι. Τα διοικητικά και νομικά θέματα τα οποία άπτονται των συναλλαγών αυτών ποτέ δεν ήταν τόσο ε, εύκολο να ξεπεραστούν όπως ε, σήμερα η, τα ποσοστά ΦΠΑ με τις διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις για τους συμβαλόμενους από πλευράς καθεστώτων και κάνοντας λόγο σε σχέση με αυτούς για, για μια τέτοια πλατφόρμα είπαν όλοι ότι μια τέτοια κοινή πλατφόρμα, ένα τέτοιο πλαίσιο θα διευκόλυνε την ζωή τους και τις συναλλαγές τους. Δεν θέλω εγώ να πω ότι θα ήταν η τέλεια λύση αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Νταϊάννα Βόλη μίλησε για ένα, μια δέσμη μέτρων, για ένα πακέτο. Η Επιτροπή μίλησε για συνοδευτικά μέτρα. Εγώ θα ήθελα αυτό το δίκαιο να είναι μια νομική πλατφόρμα μια νομική βάση για την ανάπτυξη εκείνων των πρακτικών λύσεων που θα εκπονούσαμε ώστε η ενιαία εσωτερική αγορά να λειτουργεί και να μπορεί να είναι προσπελάσιμη στους ε, χρήστες και στους συναλλασσόμενους. Ε, το όριο της φαντασίας, του εφάνταστου τρόπου δράσης θα ήταν το ε, τελικό όριο θα πρέπει εδώ να διαχέεται η πληροφορία μέσω των, του εξοπλισμού, ε, των κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε, νομίζω ότι η ίδια τα, έχουμε και τα ε, δικαιώματα επιβατών που έχουν ε, ε, διευθετηθεί και έχουν ρυθμιστεί και βλέπουμε πόσα μπορούν να γίνουν. Είναι λοιπόν ένα μέσο που θα μπορούσε να προσφέρει πρακτικές λύσεις και δυνατότητες. Πρέπει υπό όρους ελαστικότητας και διασφάλισης νομικής προστασίας με πάντα με χειροπιαστές λειτουργικές λύσεις και δυνατότητες που θα αναπτύσσονται σε συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μεταξύ των αρμόδιων για την εκπόνηση τέτοιων προτάσεων και ε, επιλογών νομικά στην, ε, ε, στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Κάποια παραδείγματα θέλω να δώσω που πιστεύω ότι είναι σημαντικά και δείχνουν σε τι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. Πρώτον, το δίκαιο αυτό θα μπορούσε να επιτρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιαδήποτε γλώσσα ο πάροχος, ο πολιτής, αντί να αφήνει τον καταναλωτή να σερφάρει για να βρει αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τη γλώσσα του στο διαδίκτυο. Αφήνοντας αυτή τη δυνατότητα ανοιχτή λοιπόν θα μπορούσε κανείς ε, σε διάφορες γλώσσες ε, να συναλλάσσεται και έτσι θα ακολουθούσαμε την τάση των ε, καταναλωτών όπως από τις επιλογές τους απορρέει. Βλέπουμε ότι 7 από 10 που απάντησαν, που απαντούν με προηγούμενη πείρα διασυνοριακά θα ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν άλλη γλώσσα στο διαδίκτυο όταν συναλλάσσονται διαδικτυακά. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να δούμε πώς θα μπορούσε το ευρωπαϊκό αυτό ε, δίκαιο να υποστηρίζει την χρήση αυτών των γλωσσικών μέσων. Διότι γνωρίζουμε ότι η γλώσσα μπορεί να είναι ένα στραγμός ή πρόσκομα. Θα έπρεπε να αφήνεται στα συνοδευτικά μέτρα να ρυθμίζουν και να αποφασίζουν πώς οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και παρουσιάζονται στον καταναλωτή. Υπάρχουν πολλές απαιτήσει ε, από πλευράς ε, του ευρωπαϊκού αυτού δικαίου και δεν πρέπει να οδηγούμε σε τρίβες. Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε τέτοιου είδους λύσεις πρέπει κινητά, στο κινητό πλαίσιο να προβληματιστούμε, να δούμε πώς αυτό θα αντανακλάται στις διάφορες συσκευές και στο διαφορετικό εξοπλισμό καθορίζοντας κάποια πράγματα και αφήνοντας κάποια άλλα εκτός. Αυτό πρέπει να επιλέξει να κάνει το δίκαιο αυτό. Και σε σχέση με την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών στους ε, καταναλωτές πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στην ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο και όχι τόσο στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των συμβαλωμένων. Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Αντανακλά το δίκαιο αυτό την ίδια την πραγματικότητα και το συσχετισμό μεταξύ των ε, ε, καταναλωτών και των παρόχων εδώ έχουμε τα ευφυή e τηλέφωνα, τα, την, τον κινητό χαρακτήρα και των υπολογιστών. Μπορούν να σερφάρουν, να, διαβάζουν, μπορούν να υποβάλουν ε, το αίτημά τους ε, διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Μπορεί να ζητήσουν κατοίκον παράδοση ή μπορεί να επιλέξουν την ε, παραλαβή από το ίδιο το μαγαζί. Εδώ πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη εξισορρόπηση σε σχέση με τις ανάγκες των καταναλωτών εξισορρόπηση των προσφορών και των πραγμάτων. Σε σχέση με την υποχρέωση, για παράδειγμα, σε σχέση με τον αγοραστή, όταν δεν θα μπορεί να παραδοθεί κατά κάποιο ε, συγκεκριμένο τρόπο ή αν θέλει να εξετάσει και να δει αν είναι το προϊόν, αν συνάδει με εκείνο το οποίο είχε παραγγείλει. Αυτού του είδους τα παιδεία, αυτή η τομή, ε, η γλώσσα, το είδος πληρωμής, ε, η πείρα των καταναλωτών και οι επιλογές και χρήσεις ε, και Φυσικά εδώ αυτά είναι θέματα τα οποία είναι μελήματα των ε, πολιτών. Θα πρέπει να μην υπάρχει κίνδυνος ε, να καταλήξει κάποιος πολιτής ε, με προσφυγή του αγοραστή σε κάποιο δικαστήριο και συνεπακολουθείς τριβές ακολουθήσουν. Σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν σε μία σύνοδο συνδιάσκεψη στο, στη Στοκχόλμη η συζήτηση είχε επικεντρωθεί σε σχέση με τις πολιτικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και είπε ο Σουηδός Υπουργό. εμείς οι υπεύθυνοι πολιτικά για την λήψη αποφάσεων πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει ο σύγχρονος εξοπλισμός και τα μέσα. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι κάνουμε με ε, την κατεύθυνση αυτή που έχουμε ακολουθήσει για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Μελίν. Στο στοχεύσαμε σε ρυθμίσεις καταναλωτών, σε διαδικασίες και ρυθμίσεις ΦΠΑ, όρους παράδοσης ή παραλαβής προϊόντος και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τους καταναλωτές, τους χρήστες, ότι ουσιαστικά να υπάρχει ένα πλαίσιο για αυτούς όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διαδικτυακές συναλλαγές να μπορούν να γίνονται σωστά. Δηλαδή να μην χρειάζεται να προβληματίζετε για άλλα πράγματα αλλά να επικεντρώνεται στο ίδιο το προϊόν, στο ίδιο το αγαθό το οποίο θέλει να επιλέξει και να μην ε, ε, αποσπάται η προσοχή του σε άλλα θέματα και αναλώνει το χρόνο του. Τώρα στη συνέχεια περνάμε στον κύριο Φραντσέσκο Σαουντόνε. Το ευρωπαϊκό αυτό δίκαιο για τις συναλλαγές παρέχει την βεβαιότητα και ασφάλεια εκείνη που αναμένουν και προσδοκούν ε, οι καταναλωτές και οι χρήστες. Δημιουργείται σαφήνεια και ευδιάκριτος ε, χαρακτήρας των όρων και προϋποθέσεων μπορούμε να αναμένουμε ότι θα επικεντρώνεται περισσότερο στα αγαθά και στα προϊόντα και να υπάρχει, να δημιουργείται νομική και, ε, ασφάλεια και βεβαιότητα ή όχι. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε εσείς κύριε Σαουντόνε παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις παρεμβάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα, το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο και είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιο είναι το δίκαιο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Και αυτό γιατί, όπως συμβαίνει συνήθως, και επικεντρώνομαι ουσιαστικά στα ζητήματα αυτά στην παρουσίασή μου, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων αποτελεί ένα προαιρετικό νομοθέτημα το οποίο θα αφορά τόσο τις συναλλαγές επιχείρησης προς καταναλωτή, όσο και τις συναλλαγές μεταξύ, επιχειρήσεων. Το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να δούμε σε σχέση με το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων είναι αν το νέο αυτό προτινόμενο νομοθέτημα επικαλύπτει ή συμπίπτει με άλλα προηγούμενα νομοθετήματα. Όσον αφορά τις συναλλαγές επιχείρησης προς καταναλωτή, θεωρούμε ότι υπάρχει επικάλυψη με την Οδηγία 83 κάθος 2011 και όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων υπάρχει επικάλυψη με τη Σύμβαση της Βιέννης. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο ως δικηγόροι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί ως συνήθως καλούμαστε εμείς να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το δίκαιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Μέσω της παρουσίασης αυτής θέλουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μειωθούν στο σημείο του δυνατού όλες αυτές οι γκρίζες ζώνες οι οποίες παραμένουν στο νομικό πλαίσιο της πρότασης αυτής. Εξετάζοντας τις επικαλύψεις που υπάρχουν στις συναλλαγές επιχειρήσεων καταναλωτών, αν δούμε το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων και την Οδηγία 83 του 2011, βλέπουμε ότι το πεδίο εφαρμογή είναι συναφέ, συμπίπτη. Η οδηγία αναφέρεται σε οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, ενώ το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πωλήσεων αναφέρεται στι διασυνοριακέ συμβάσει μεταξύ πολιτών και καταναλωτών. Το πεδίο εφαρμογή των δύο αυτών νομοθετημάτων καταδεικνύουν ότι οι περισσότερε συναλλαγέ και συμβάσει που καλύπτονται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων ήδη καλύπτονται από την οδηγία. Και ουσιαστικά ότι η ιδιοποιώς διαφορά είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές μόνο και τίποτα άλλο. Η πρόταση λοιπόν για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων έχει πολλές κοινέ διατάξεις με την υφιστάμενη οδηγία, όπως για παράδειγμα οι απαιτήσει πληροφόρησης, το δικαίωμα επαναχώρησης, οι διατάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την παράδοση των αγαθών. Σε όλους αυτούς τους τομείς θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνταχθεί η πρόταση κατά τέτοιον τρόπο, προκειμένου πραγματικά να αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των Πωλήσεων σε σχέση με την οδηγία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τι επιχειρήσει αλλά και για του καταναλωτέ. Μία άλλη επικάλυψη που έχουμε εντοπίσει είναι αυτή που έχει να κάνει με τα κοινά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην Σύμβαση της Βιέννης και στο Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Οι διασυνοριακές συναλλαγές καλύπτονται από τη Σύμβαση της Βιέννης, από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Πέρα από το κοινό πεδίο εφαρμογή, τόσο η ΣΥΣΛ όσο και η Συνθήκη της Βιέννης ουσιαστικά είναι προαιρετικά συστήματα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα συμβαλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν και από τα δύο αυτά νομοθετήματα. Αυτό το δικαίωμα αυτεξαίρεσης λοιπόν που προβλέπεται από τη Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών παρουσιάζεται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βλέπουμε ότι ε, η συνθήκη της Βιέννης ασχολείται με τις εμπορικές συμβάσεις, ρυθμίζει εμπορικές συμβάσεις. Ένα 90% των συμβάσεων αυτών προβλέπουν μια ρήτρα διετησίας. Από την άλλη προβλέπεται η δυνατότητα opt-out και από τα δύο νομοθετήματα και το επίπεδο opt-out είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν προτού ολοκληρώσουμε τον κανονισμό για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων να δούμε ακριβώ τι συμβαίνει με το CISG, τι συμβαίνει με τη συνθήκη τη Βιέννη. Για ποιο λόγο τα περισσότερα συμβαλόμενα μέρη αποφασίζουν να αυτεξαιρεθούν από τη συνθήκη τη Βιέννη. Αν λύσουμε το ζήτημα αυτό θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την ίδια αντιμετώπιση και για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Για ποιο λόγο όμως πάρα πολλά συμβαλώμενα μέρη επιλέγουν να αυτεξαιρεθούν. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει οι οποίε αποφασίσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζουν ακριβώ πώ λειτουργεί η συνθήκη τη Βιέννη, γιατί υπάρχουν κάποιε τυποποιημένε συμβάσει οι οποίε δεν επιθυμούν να υιοθετήσουν και γιατί υπάρχουν και κάποιε συγκεκριμένε ανησυχίε. Ένα από τα δύναμα σημεία τη συνθήκη τη Βιέννη είναι ότι δεν καλύπτει τον συνολικό κύκλο ζωή τη σύμβαση. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν κανόνε όσον αφορά την έλλειψη συνένεση, δεν υπάρχουν κανόνε όσον αφορά τα καθήκοντα ενημέρωση και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε όσον αφορά τι γενικέ ρήτρε. Αυτή η ατέλεια, αυτή η έλλειψη πληρότητας δημιουργεί τελικά ένα κατακαιρματισμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά επιμέρους μέρη συμβάσεων, τα οποία καταλήγουν τελικά να καλύπτονται μόνο από τεχνική νομοθεσία στο τέλος και όχι από το CISG. Επίσης, Κατά αυτόν τον τρόπο μια σύμβαση μπορεί να υπόκειται σε πολλά διαφορετικά νομοθετήματα, από τη μια στη Διεθνή Σύμβαση και από την άλλη σε εθνικά συστήματα. Ο κατακαιρματισμό αυτό δημιουργεί όμω πολυπλοκότητα, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούν βέβαια οι επιχειρήσεις. Ποια είναι τώρα τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από την κατάσταση αυτή. Ο φόβο του κατακαιρματισμού και της πολυπλοκότητας οδηγεί τελικά σε αυξημένα επίπεδα opt-out. Οι περισσότερε επιχειρήσει προτιμούν να έχουν μία και μοναδική νομοθεσία. Συντοποιούμε λοιπόν ότι η πληρότητα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου ένα νέο σύστημα να, είναι, να στεφτεί με επιτυχία. Τώρα, από πρακτικής πλευράς, πρέπει να εξετάσουμε και ποια είναι η επίπτωση των τυποποιημένων συμβάσεων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει πάρα πολλούς πόρους στο να δημιουργήσουν κάποιες πρότυπες συμβάσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους. Τις περισσότερες φορές οι συμβάσεις αυτές εξαιρούν την εφαρμογή της συνθήκης της Βιέννης. Και πιστεύουμε βέβαια ότι στο μέλλον μπορεί οι συμβάσεις αυτές να μην χρησιμοποιούν καν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων, το οποίο θα είναι και προαιρετικό μέσο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες θα αποφασίσουν να μην επανασχεδιάσουν τις πρότυπες συμβάσεις τους προκειμένου αυτές να συνάδουν με το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Τώρα, θα πρέπει να αφαιρθούμε επίσης στη σχέση που υπάρχει μεταξύ κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων και της προστασίας των καταναλωτών. Οι περισσότερες ε, διατάξεις του προτινόμενου καονισμού θέλουν να πετύχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους αδύναμους και τους δυνατούς συμβαλόμενους. Θεωρούμε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν επιτυχάνεται όταν η συναλλαγή είναι μεταξύ επιχειρήσεων. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αναλύσουμε εδώ πέρα περισσότερο την κατάσταση και να δούμε τελικά αν τελικά με τον προτινόμενο καονισμό που απλοποιούμε ή όχι τα πράγματα. Πραγματικά χρειαζόμαστε τη νέα αυτή νομοθεσία στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και εγώ θα μπορούσα να αφαιρθώ αυτή τη στιγμή σε δύο σενάρια. Σε μια συναλλαγή ανάμεσα σε μια μεγάλη επιχείρηση και μια μικρομεσαία επιχείρηση ή σε μια συναλλαγή μεταξύ δύο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας αναλύσουμε τα δύο αυτά σενάρια. Στην πρώτη περίπτωση, στη συναλλαγή ανάμεσα στην ε, μεγάλη επιχείρηση και τη μικρομεσαία επιχείρηση, βλέπουμε ότι υπάρχει όντως μία ανισορροπία. Και ότι ενδεχομένω εδώ πέρα όντω να δικαιολογείται ένα κανόνα που να προστατεύει το πιο αδύναμο μέλο. Θα αποδέχονταν όμω οι μεγάλε επιχειρήσει να υιοθετήσουν μια νομοθεσία η οποία θα προστατεύει τον αντισυμβαλόμενο, τον πιο αδύναμο αντισυμβαλόμενο. Ας πάρουμε τώρα το δεύτερο σενάριο. Συναλλαγή μεταξύ δύο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποια ανισορροπία. Δεν υπάρχει ένας δυνατός και ένας αδύναμος συμβαλόμενος. Στην περίπτωση αυτή, το αυξημένο επίπεδο προστασίας για το ένα μέρος τελικά της σύμβασης ουσιαστικά δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Εν κατακλείδη λοιπόν, μπορώ να πω τα ακόλουθα. Ο προτινόμενος κανονισμός ουσιαστικά επικαλύπτει την οδηγία η οποία ήδη ισχύει και ο κανονισμός ε, αυτός θα πρέπει να εξεταστεί ακόμα περισσότερο για να δούμε τελικά ποια είναι η επίπτωση που ήδη υπάρχει από την οδηγία και πώς θα μπορούσαμε από τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από την οδηγία να βελτιώσουμε περισσότερο από τον καονισμό. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες νομικού περιεχομένου και οι καταναλωτές επίσης θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες πανευρωπαϊκά όσον αφορά τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και πώλησης. Προετοιμαζόμενοι λοιπόν για την νέα αυτή νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά. Ξέρετε ότι οι δικηγόροι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε θέση να συμβουλεύσουν τους πελάτες για τα υπέρ και τα κατά της χρήσης αυτού του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των Πολίσεων ακόμα και αν η χρήση του παραμένει προαιρετική. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Σιαουντώνε για τα όσα μας ε, εκθέσατε χωρίς να θέλω τώρα να πω ότι είπατε κάτι να το βάλω στο, στα όσα αναφέρατε θα μπορούσε κανείς να αποκομίσει την εντύπωση το κοινό αυτό ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών βρίσκεται σε αντιδιαστολή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως ισχύουν σήμερα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί, αλλά παραμένει το ερώτημα. Εκκρεμεί και αναμένει απάντηση. Περνάμε στον επόμενο αγορητή. Είναι ενδεδειγμένο το ευρωπαϊκό αυτό συναλλαγών ώστε να διασφαλίζει την βέλτιστη προστασία καταναλωτών είναι ένα ευρύ πλαίσιο και πρέπει να δούμε όλες αυτές τις πτυχές. Όλες οι ελπίδες και οι προσδοκίες μπορούν να υλοποιηθούν ή πρέπει κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα να επικεντρωθούμε και σε αυτά να ε, εμβαθύνουμε. Δεν θέλω εγώ να προδικάσω, σας δίνω τον λόγο κύριε Κρίγκερ να μας τα πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα γερμανικά. Η δική μου προσέγγιση επηρεάζεται από τα βιώματα που είχα ως ε, επικεφαλής ε, του Κέντρου Προστασίας ε, Καταναλωτών, του Κέντρου Καταναλωτών, Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη Γερμανία. Δουλειά μας είναι τα προτερήματα, να ενημερώσουμε για τα προτερήματα που υπάρχουν στην ενιαία εσωτερική αγορά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτή την αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά και συμμετέχουμε όταν υπάρχουν τριβές και προβλήματα στην επιδιαιτησία μέσα στο πλαίσιο του ε, δικτύου είχαμε <clears throat> περίπου 9.200 τέτοιες περιπτώσεις και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών συμμετείχε με πάνω από 30% στις δράσεις και από κοινού με τους Γάλλους συναδέφους που συστεγαζόμαστε είχαμε περίπου το ίμιση των περιπτώσεων στις οποίες ε, είχαμε εμπλακεί. Κάνω λόγο λοιπόν για την διασυνοριακή ε, πτυχή των συναλλαγών υπό το πρίσμα των χρηστών, των καταναλωτών. Μπορεί κανείς να πει ότι ένα κοινό δίκαιο είναι ενδεδειγμένο ώστε να αρθούν τα εμπόδια για την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Αν μέσω αυτής της οδού, αυτής της πορείας, μέσω της προαιρετικής δυνατότητας ένταξης των 28 αστικών ε, νομοθεσιών αν έτσι πρακτικά μπορεί η πρόσβαση ε, των καταναλωτών να διευκολύνεται και μάλιστα με μακροπρόθεσμο χρονοορίζοντα και έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις. Πρώτη επιφύλαξη ξεκινάμε ήδη με το ότι στην πρακτική εφαρμογή το θέμα του εφαρμοστέου δικαίου κατά κανόνα έχει υποδέστερο ρόλο όταν πρόκειται για τα εμπόδια, για παράδειγμα, ή τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν ε, οι καταναλωτές, οι χρήστες ε, που θέλουν κάτι να αγοράσουν, είναι ουσιαστικά τα προσκόμματα τα γλωσσικά είναι η απουσία της προθυμίας ε, του παρόχου να παρέχει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά αυτά σε μια συγκεκριμένη χώρα και η μη δεδομένη προθυμία να αποδέχονται πιστοτικές κάρτες ε, στις συναλλαγές αυτές. Αυτά όλα μπορέσαμε να τα διαπιστώσουμε σε όλες τις δράσεις που κάναμε. Και επιπλέον ο κατακαιρματισμός του δικαίου είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο σε σχέση με τα προσκόμματα και εμπόδια στις διασυνοριακές αυτές συναλλαγές. Πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε ότι ιδιαίτερα με τις τηλεαγορές και από πλευράς της συναδέφου προαναφέρθηκε αυτό, ένα πολύ μεγάλο μέρος των διασυνοριακών ε, συναλλαγών είναι τέτοιου είδους τηλεαγορές. Κατά κανόνα, ο πάροχος, εκείνος που προσφέρει με τις διαφημίσεις του και την διάχυση ε, στοιχείων για αυτό το προϊόν, από την άλλη πλευρά ε, τα συνδέει όλα αυτά με το οικείο για τον χρήστη δικό του νομικό πλαίσιο και από τότε που έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Σεπτεμβρίου από πλευρά νομολογία στι περισσότερε περιπτώσει θα μπορούσε να επιλεγεί αυτό το ε, πλαίσιο ω ισχύον πλαίσιο και επιπλέον έχουμε και τη σημασία των γνώσεων που έχουν για τα δικαιώματά του οι καταναλωτέ, που ιδιαίτερα στη διασυνοριακή συναλλαγή έχουν υποδέστερο ρόλο όλα αυτά τα δικαιώματα και η προστασία τους αν λάβουμε υπόψη ότι πληρώνει πρώτα ο ε, αγοραστής και μετά παίρνει το εμπόρευμα, το αγαθό. Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο λοιπόν, η εμπιστοσύνη όσον αφορά τον προσφέροντα ή τον πάροχο. Χωρίς εμπιστοσύνη προς τον πάροχο ή τον προσφέροντα δεν μπορεί να υπάρξει η ορίμανση μιας συναλλαγής, η επίτευξη η επιτευξη συναλλαγη Και το θέμα του δικαίου που θα ισχύει μόνο τότε στη συνέχεια μπορεί να εξεταστεί. Όταν δηλαδή ε, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και πρέπει τότε να διερωτηθεί ο καταναλωτής, καταναλωτής πού θα υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου και ποιο δίκαιο θα ισχύει. Έχουμε λοιπόν σημαντικές αμφιβολίες αν αυτό το δίκαιο συναλλαγών την πρόσβαση στις διασυνοριακές συναλλαγές τη διευκολύνει ε, ουσιοδός ή όχι. Και τώρα έχουμε και ένα πρόσθετο στοιχείο. Φοβόμαστε ότι αυτή η παράλληλη συνύπαρξη δύο διαφορετικών νομικών καθεστώτων θα μπορούσε να συνεισφέρει στο ότι ακριβώς η επιλογή του ευρωπαϊκού δικαίου συναλλαγών που την βρίσκουμε θετική ως προσέγγιση αλλά που οδηγεί στο, θα μπορούσε να οδηγήσει να πόσχουν από αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο οι καταναλωτές, οι χρήστες η πείρα μας δείχνει ότι όταν έχουμε προαιρετικά την επιλογή ενός καθεστώτος, ακόμα και ενήμεροι και πληροφορημένοι αγοραστές ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, ένα τέτοιο, ας το πω ε, στοιχείο και προτιμούν τα οικία καθεστώτα και ξεκινούμε με την διαφοροποίηση μεταξύ εγγυήσεων και παροχή περίοδου εγγύησης και που δημιουργούνται οι πρώτες δυσκολίες. Υπό αυτό το σκηνικό δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αν λέγαμε σε κάποιον καταναλωτή ότι ξέρεις έχεις την επιλογή μεταξύ αυτής και της άλλης ε, ε, νομικής τάξης πραγμάτων ότι τότε θα μπορούσε αυτός να επιλέξει το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο συναλλαγών. Θα ήθελα να πω και κάτι για τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις σε σχέση με τον τύπο όταν πρωτογνωρίστηκε αυτό, αυτή η προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την ενημέρωση τύπου αναφέρθηκε ότι θα υπάρχει η επιλογή να επιλέγει κανείς ένα φιλικό προς το χρήστη πλαίσιο κάνοντας ένα κλικ με το ποντίκι μόνο στο ε, διαδίκτυο ηλεκτρονικά σε σχέση με τα δικαιώματα που θα είχε από πλευράς αυτού του δικαίου. Κοιτάζοντας το αυτό ο καταναλωτής πρέπει να πω δεν έχει ακριβώς την επιλογή μεταξύ του οικίου δικαίου το οποίο γνωρίζει και του νέου συμβατικού δικαίου για τις συναλλαγές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έμπορος είναι εκείνος ο οποίος έχει την επιλογή να θέσει τον αγοραστή ενώπιον της επιλογής ή να επιλέξει το, ε, το πλαίσιο το οποίο του προτείνεται είναι απόσχεια από αυτή τη συναλλαγή. Και κατά τούτο λοιπόν είναι ο ιτημένος εντός εισαγωγικών ο αγοραστής. Δεν μπορεί ο ίδιος να επιλέξει, του επιβάλλεται ένα καθεστώς. Και δεν υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρξει σύναψη μιας ευρωπαϊκής σύμβασης αγοράς. Και αυτό θα μπορούσε να γινόταν με ένα κλικ με το ποντίκι. Και έτσι αντιμετωπίζει μια κατάσταση που δεν μπορεί να την ξεπεράσει ο ε, αγοραστής ίσως και αμφότερη διότι δεν είναι ένα πρότυπο σύμβασης ή συναλλαγής ε, αυτή η αγορά όπου δηλαδή οι όροι θα ήταν παντού οι ίδιοι για όλους και όπου θα ίσχυε μια τέτοια, ένα τέτοιο πρότυπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βλέπουμε ότι ο επιχειρηματίας έχει ένα ε, ε, όργανο, ένα μέσο αστικού δικαίου, χαρακτήρα αστικού δικαίου στα χέρια του που μπορεί να το προσαρμόσει, να το τροποποιήσει και αυτό πάλι οδηγεί τον επιχειρηματία να χρειάζεται νομομαθείς ή νομοσυμβούλους για να προχωρήσει. Εδώ πιθανόν καταναλωτές θα μπορούσαν να δεχθούν ένα τέτοιο ευρωπαϊκό δίκαιο αν υπήρχε η επικοινωνία προς αυτούς και τους εξηγεί ότι τότε θα βρισκόντουσαν σε καλύτερη θέση από ό,τι προηγούμενα σε σχέση με ένα εθνικό καθεστώς. Αλλά φοβούμε και αυτός ο φόβος προαναφέρθηκε ότι αυτό δεν θα, μπορούσε ε, να, δεν θα μπορούσαμε να το εγγυηθούμε σε όλες τις περιπτώσεις και θα υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις αρνητικές όπου θα μπορούσε κανείς να αποδείξει ότι θα υπρόκειτο και για μια αρνητική διαφήμιση. Πολλές φορές ε, ε, θα μπορούσε κανείς να φοβηθεί ότι αν κάτι κάτι κάπου ε, φοβάται ο αγοραστής ε, ως μειονεκτικό ή αρνητικό για εκείνον θα τον έκανε να μην επιλέξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο συναλλαγών. Και ένα επιπλέον στοιχείο υπάρχει εδώ. Η συμβατική ελευθερία, η ελευθερία της ε, σύναψης συμβάσεων. Δεν θα μπορούσε να αποκλείει κανείς ότι θα εξακολουθούσαν να παρέχονται αυτές ε, οι ε, διευκολύνσεις σε σχέση με το εθνικό πλαίσιο συναλλαγών. Ιδιαίτερα για παράδειγμα για το κόστος μεταφορών που είναι ένα ε, μείζον εμπόδιο για τους εμπόρους σε σχέση με την παράδοση αγορών αγαθών στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν πολύ μεγάλες προσδοκίες να δημιουργηθούν που δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στο τέλος και να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κρίγκερ. Αρκετά στοιχεία είχαμε εδώ που ακούσαμε που τα συζητήσαμε και την τελευταία εβδομάδα και με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και με τους ε, Ευρωβουλευτές. Ακούγοντας τώρα την δήλωση της κυρίας Μελίν και αθρίζοντας και αυτήν στο σύνολο, η εντύπωσή μου είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ολοκληρώσαμε ακόμα, ότι υπάρχει το ένα ή άλλο σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί, αλλά υπάρχει επίσης και ανάγκη. Ανάγκη και ζήτηση. Ζήτηση ακριβώς στο online για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κυρία Μελίνος, εκπρόσωπος ε, του εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, μας δείχνει μια ε, κατεύθυνση. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή κατεύθυνση όλοι όμως. Αδειμονώ να ακούσω προς τα που θα κατευθυνθούμε. Έχουν ζητήσει αρκετοί τον λόγο. Κάποιες παρεμβάσεις έχουμε. Ίσως οι τοποθετήσεις του πρώτου μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις παρεμβάσεις του δεύτερου πάνελ σε μια συνολική εικόνα που θα αποκομίσουμε. Δήλωση ή ερώτηση, δεν είμαι βέβαιος περί τίνος πρόκειται, ο κύριος Πιότρο Τσιντάσκι, συνάδελφος από την Γερουσία της Πολωνίας. Σας δίνω τον λόγο κύριε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πρέπει να πω αυτή η συζήτηση. Και εγώ ο ίδιος προσωπικά είμαι πρόεδρος της ε, Νομικής Επιτροπής ε, της ε, ΣΕΜ στη, στη Βουλή της Πολωνίας. Ε, επί δεκαετίες ε, ήμουν δικηγόρος και τα προβλήματα της νομικής, της άσκησης ε, του, πρακτικής εφαρμογής του δικαίου είναι κάτι που παρακολουθώ του σύνεγγυς. Σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει μια επιφύλαξη που διατυπώθηκε και ακούστηκε. Δεν θα ήθελα η συζήτηση επ' αυτού να περιοριστεί και να πούμε ότι όσον αφορά την Πολωνία η έγκριση, η αποδοχή αυτού του μέσου, του ευρωπαϊκού ε, μέσου, του ευρωπαϊκού χαρακτήρα, το υποστηρίζουμε κοινέ προδιαγραφές και διατάξεις ε, για τις συναλλαγές για ένα εμπορικό δίκαιο που θα ίσχυε σε όλες τις ε, χώρες μέλη ώστε η έγκριση αυτού του μέσου και η αποδοχή του, η θέσπιση του και ακριβώς από νομικής πλευράς υπομορφή κανονισμού θα έπρεπε να γίνει η έγκριση αυτού του μέσου. Και ε, υποστηρίζουμε και το πλαίσιο της ε, εθελοντικής συμμετοχής, της προαιρετικής συμμετοχής των συμβαλωμένων. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σε ένα ερώτημα. Σε ένα ερώτημα το οποίο απορρέει και από την παρουσίαση του κυρίου καθηγητού Σιμονίδη που ακούσαμε πιο πριν, Σιμεωνίδη, του εκπροσώπου της Κυπριακής Προεδρίας. Τι είπε ο κύριος Σιμεών Σιμεωνίδης. Είπε ότι εδώ πρόκειται για ένα θέμα που δεν μπορεί να διευθετηθεί εν μια στιγμή. Χρειάζεται μια χρονική προοπτική και αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ένα χρονικό πλαίσιο πιο μεγαλόπνο. Δεκαετία για παράδειγμα μπορεί να είναι αυτό το χρονικό πλαίσιο. Βλέπουμε ήδη τα προβλήματα και αυτό είναι θετικό. Ανοιχνεύουμε προβλήματα τα οποία επί πρακτικής ε, μορφής σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να επιληθούν. Εγώ θα εκφραζόμουν υπέρ του ότι η πρόταση του καθηγητού Στάουντεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή ο οποίος καθηγητής Στάουντεν Μάιο τι ανέφερε. Ανέφερε ότι ε, έκανε ε, μια παρατήρηση για τα σχόλια για σχολιασμό. Ακούσαμε επίσης και την τοποθέτηση του καθηγητού Φόγενάουερ, ο οποίος μίλησε για το δίλημα, αιώνιο δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αν ο αποδέκτης αυτής της ρύθμισης είναι η νομομαθείς ή αν είναι οι επιχειρηματίες, οι χρήστες, οι καταναλωτές. Το σχόλιο όμως αυτό συνενώνει αυτές τις δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Ένα σχόλιο ερμηνευτικό όμως που πρέπει να είναι να βασίζεται σε πολυετή πείρα και πρακτική όσον αφορά την ομολογία των δικαστηρίων για παράδειγμα και μόνο με τέτοια προσαρμογή και πρακτική έχει πρακτική αξία ένα τέτοιο σχόλιο. Σας, ευχαριστούμε θερμά. Παράλληλα με την στεναρή αυτή τοποθέτηση είχαμε και ερώτηση προς τον καθηγητή κύριο Σημεωνίδη θα ήθελα να ακολουθήσω αυτή τη σειρά και επιτρέψτε μου να σας δώσω τον λόγο στο τέλος, αντιστρέφοντας τη σειρά, διότι και αυτό το ερώτημα θα πρέπει να παραμείνει. Συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις με τη σειρά τους. Αλτάβα Λαβάλ από το, την Ισπανική Γερουσία, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το έργο των εισηγητών που που και σήμερα στην εξαντλητική αυτή ημερίδα και περιεκτική μερίδα καθώς και για τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλουν στις μελέτες τους σε σχέση με μια κοινή προοπτική, ευρωπαϊκή προοπτική για τη ρύθμιση των συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είμαι αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης στην ε, ε, Ισπανική Γερουσία και θεωρώ ότι πολύ καλά μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια ρύθμιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα για τι συναλλαγέ για να προσεγγίσουμε τα θέματα των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτά. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι τέσσερις οι ευρωπαϊκές ελευθερίες. Ελευθερία κυκλοφορίας των ατόμων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Και με αυτή την έγκριση, με την έγκριση αυτού του μέσου θα καταφέρουμε να πείσουμε, να δείξουμε ότι έχουμε πιστεί για τη σημασία ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία αυτών των αγαθών. Είναι λοιπόν ένα βήμα κέρια σημασία, θεμελιώδου σημασία ε, για να πετύχουμε την ρύθμιση θεμάτων της, ε, του συμβατικού δικαίου, τη σύναψη ε, συμβάσεων. Κάποια ερωτήματα απορρέουν όμω, κάποια ερωτήματα τα οποία απορρέουν από τι παρεμβάσει και που στη συνέχεια θα παρουσιάσω. Προβλέπεται προαιρετικό χαρακτήρα αυτού του μέσου για τι επιχειρήσει, μικρομεσαίε επιχειρήσει και για χρήστε που προαιρετικά θα μπορούν να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο. Επίση, Επίσης και οι δημόσιες αρχές και διοικήσεις, το κράτος μέσω οποιασδήποτε ε, υπηρεσίας του, είτε είναι διοικητικού χαρακτήρα, είτε θεσμικού χαρακτήρα, είτε συλλογικού χαρακτήρα, θα μπορούσε εθελοντικά, προαιρετικά το κράτος να ενταχθεί σε ένα τέτοιο μέσο, μια και όλο και περισσότερο συμμετέχει στην ε, ρύθμιση τέτοιου είδους συμβάσεων, όχι μόνο διοικητικών συμβάσεων που είναι χαρακτηριστικές ε, του ε, διοικητικού χαρακτήρα, αλλά και συμβατικού χαρακτήρα αγοραπολισιών και ίσως λόγω επαγγέλματος θέτω την δικονομική πλευρά του θέματος στο επίκεντρο. Δικονομικά δεν είδα να ρυθμίζεται κάτι από αυτό το μέτρο. Όντας εθελοντικού χαρακτήρα προαιρετικό, κατανοώ ότι δικονομικά η εφαρμογή αυτών των θεμάτων και όσον αφορά τις διατάξεις θα απομένει στην ε, διακριτική ευχέρεια των συμβαλωμένων. Ελεύθερα θα αποφασίζουν τα συμβαλώμενα μέρη προς ποιο δικαστή θα προσφύγουν σε περίπτωση ύπαρξης ε, προβλήματος. Αν δεν υπάρχει καθορισμός ενός τέτοιου μέσου, ποιος είναι ο δικαστής ο οποίος ε, θα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει και θα επιληφθεί τη ρυθμίσεως ενός τέτοιου προβλήματος όταν και αν υπάρξει ένα τέτοιο πρόβλημα. Κατανοώ ότι θα εφαρμόζονται εδώ οι αρχές του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το μέσο κάτι αναφέρει, η πρόταση αναφέρει κάτι σχετικά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση αυτού του ερωτήματος. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ θερμά. Και εδώ πάλι τα ερωτήματα αυτά με τη σειρά θα τα πάρουμε και θα τα διαβιβάσουμε στους ειδικού για να τα απαντήσουν στη συνέχεια. Ιδιαίτερα για το δικονομικό δίκαιο. Αλλά ο επόμενος αγορητής ε, όσον αφορά την συνέχεια Λέον Γκλόντεν από το Λουξεμβούργο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βουλευτής και ε, συμμετέχω στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Αν δούμε την κατάσταση στο Λουξεμβούργο, βλέπουμε ότι ένα 52% των παραγγελιών που γίνονται μέσω του ίντερνετ από το Λουξεμβούργο προς το εξωτερικό δεν ολοκληρώνουν τελικά γιατί αυτές οι εταιρείες στο εξωτερικό δεν θέλουν να ε, επιβάλλουν το ε, δίκαιο του Λουξεμβούργου, να συμμορφωθούν με το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Έχουμε πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο. Έχουμε 165.000 ανθρώπους οι οποίοι διέρχονται τα σύνορα του Λουξεμβούργου προκειμένου να εργαστούν από το Βέλγιο, την Γαλλία ή τη Γερμανία στο Λουξεμβούργο και γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι τους. Επομένως, το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου είναι σαφώς ε, υπέρ της ε, πρότασης αυτής. εξετάζουμε συγκεκριμένα κεφάλαια του σχεδίου κανονισμού στη δική μας την Επιτροπή, στο δικό μου το Κοινοβούλιο. Προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν. Ένα σημείο στο οποίο χωλαίνει κάπως η πρόταση είναι στο ότι, στο, στο ότι επικεντρώνεται πάρα πολύ στην προστασία των καταναλωτών. Πάρα πολλοί ομιλητέ το είπαν σήμερα, στη σημερινή μα συνεδρίαση, ότι έχουμε ήδη ένα δίκαιο το οποίο προστατεύει πάρα πολύ τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο επί τα στεπιμέρους κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και την προστασία του ίδιου του εμπορίου. Εν τέλει θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βγει μόνο κερδισμένη από τον νέο αυτό κανονισμό όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων, ιδίω στην περίοδο αυτή της κρίσης που διανύουμε. Θεωρώ ότι ε, πρέπει να προωθήσουμε και αυτό το επιχείρημα αύξηση ανταγωνιστικότητα το οποίο θα έρθει μέσω αυτού του δικαίου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αρκετού που θέλουν να παρέμουν στη συνέχεια. Επόμενος, ο Λέορδο Μπόνε. Και μετά ο συνάδελφος Λένε. Μετά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Σιμεωνίδη για να απαντήσει αν επιθυμεί αυτή την ερώτηση και στον καθηγητή Σούλτ για τις ε, ερωτήσεις αυτές που διατυπώθηκαν. Μπορούν τέτοιου είδους συμβάσεις να χρησιμοποιηθούν ως δυνατότητες και από το κράτος ή τις ε, διοικητικές αρχές και μετά θα ολοκληρώσουμε με τις παρεμβάσεις των εισηγητών και θα περάσουμε στον κύριο Νεράντζη Τώρα και Ζέλαφελτ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή, ο κύριος Στάουντερ Μάιερ ζήτησε και εκείνο να παρέμβει. Όποιος θέλει να παρέμβει μπορεί να το γνωστοποιήσει. Με αυτή τη σειρά όμως θα πρότεινα να ακολουθήσουμε τη σειρά των παρεμβάσεων. Επόμενος ο Λόρδος Μπόουνες παρακαλώ. Thank uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε δύο ερωτήματα θα ήθελα να αφαιρθώ απευθυνόμενο στον κύριο Μάιερ. Ακούσαμε σήμερα το απόγευμα εμπειρογνώμονες αλλά και πολιτικούς οι οποίοι εξέφρασαν κάποιους ενδιασμούς για διάφορα στοιχεία της πρότασης αυτής, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές. Υπόθηκε ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε το διασνοριακό εμπόριο, αν δεν ικανοποιημένοι όσοι συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τότε δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι στόχοι όμως ουσιαστικά είναι καλοπροαίρετοι παγκοσμίω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χαθεί, αν η υφιστάμενη πρόταση ως έχει αποτελέσει τελικά σχέδιο κανονισμού και δεν τροποποιηθεί. Απευθύνω λοιπόν ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη ζήτηση που έγινε εδώ πέρα σήμερα το απόγευμα. Θα αποκομίσουν κάποια διδάγματα τελικά και θα προσπαθήσουν να εστιάσουν περισσότερο την πρόταση αυτή σε συγκεκριμένα σημεία, να είναι πιο καλαστιασμένη δηλαδή. Και μια δεύτερη παρατήρηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η δική του συστάση όσον αφορά το ζήτημα της νομικής βάσης, ζήτημα το οποίο έχουν θίξει πολλοί παρεμβαίνοντες και κατά τη διάρκεια τη σημερινής συνεδρία, αλλά και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Επόμενος, ο κύριος Κλάους Χανερλένε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Θα ήθελα, μια και μια ολόκληρη σειρά παρεμβάσεων έγιναν, υπό το πρίσμα του εισηγητού και υπό το πρίσμα και των δύο συνεισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να παραστεί ο κύριο Μπερλιγκουέρ, έχει ανηλυμένη υποχρέωση κατεπήγοντο χαρακτήρα και πρέπει να βρίσκεται στη Ρώμη. Αλλά και υπό το πρίσμα του ενό εισηγητού θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία διαδραμάτισαν ένα ρόλο στη συζήτηση. Αρχίζω με την έννοια νομική κατάσταση των πραγμάτων, νομική βάση. Ομολογώ αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε σε βάθο. Το κάναμε ήδη εμεί εσωτερικά στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Η εκκίνηση είναι ότι και οι τρει νομικέ υπηρεσίε και των τριών θεσμικών οργάνων. Η νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου κατέληξαν ομόφωνα στο αποτέλεσμα ότι η σωστή νομική βάση είναι το άρθρο 114. Επιχειρηματολογούν και λένε ότι το άρθρο 152 είναι μια ε, συνεπικουρική νομική βάση που μόνο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν χρησιμοποιηθεί το άρθρο 114. Συμφωνούν και συμπίπτουν οι τρει νομικέ υπηρεσίε. και παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι δεν είναι πιθανό ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα αποφασίσει αποφασίσει διαφορετικά από ό,τι συνιστούν και οι τρεις νομικές υπηρεσίες. Είναι ένα γεγονός από το οποίο δεν μπορούμε να απόσχουμε. Είναι γεγονός από αυτό το σημείο θα πρέπει να κινήσουμε για την διεξαγωγή της περαιτέρω συζήτησης. Συνεπικουρικότητα και επ' αυτού κάποιες δύο ε, παρατηρήσεις. Έχουμε μια πρόταση ενώπιόν μας που είναι το πιο ήπιο μέσο ώστε σε σχέση με την επέμβαση στην ε, ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο να μην επέμβουμε περισσότερο. Δεν πρόκειται εδώ για θέματα εναρμονισμού. Πρόκειται αποκλειστικά για διασυνοριακές ε, τέτοιες ε, υποθέσεις επικουρικά, ε, εθελοντικά να μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο συμπληρωματικό μέσο. Το πιο ήπιο από πλευράς νομικού χαρακτήρα μέσο όσον αφορά τις εθνικές, τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα για τη ρύθμιση τέτοιων θεμάτων εθνικά. Και αυτό δείχνει γιατί έχουμε μια νομική κατάσταση σύμφωνα με την οποία το εθνικό δίκαιο συνήθως έχει ανέβοντα ρόλο. Και εδώ βλέπουμε την ευρωπαϊκή διάσταση σε σχέση με τις διατάξεις της Ρώμης 1. Αυτή η ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τους ε, κανόνες και την ε, παρέκκληση αυτή είναι μια επίπτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν το επιχείρημα της επικουρικότητας δεν μπορεί να είναι πιστικό και το αναφέρω αυτό είναι η επικρατούσα άποψη στην Επιτροπή Νομικών ε, υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερο θέμα, αν ο πλήρη εναρμονισμό θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη πορεία προ το μέλλον. Συμμερίζομαι την άποψη. Ο πλήρη εναρμονισμό στην Ευρώπη θα ήταν η σωστή πορεία. Αυτό θα είχε για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει και την οικονομία θα ήταν η καλύτερη πορεία. Αυτό είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσει και οι οικονομικοί κύκλοι ζητούν τον πλήρη εναρμονισμό. Το πρόβλημα όμω ποιο είναι. Πολιτικά δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Δεν είναι εφικτό. Και για, την ελίπουσα, ε, για τον ελίποντα πλήρη εναρμονισμό είναι η οδηγία περί ε, συμβατικών υποχρεώσεων. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι μετά από σύσταση των πραγματογνωμόνων προβλέπεται και πρέπει να ακολουθηθεί ο πλήρης εναρμονισμός και στα δύο σώματα και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για πολλούς λόγους απέτυχε αυτό το εγχείρημα και δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Είναι σαφές ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει και ε, σε σχέση με το κάστοτε ανώτερο ε, επίπεδο προστασίας από πλευρά των κρατών μελών μέσα στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού που θα έπρεπε να είχε εξευρεθεί και μεμονωμένα για όλους ε, τους καταναλωτές και για όσους συνάπτουν προκύπτουν τέτοιες συμβάσεις ε, εσωτερικά ε, ε, στο εθνικό πλαίσιο και για τους άλλους που συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις ευρωπαϊκά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες διακριτικές αρνητικές αντιμετωπίσεις. Αν όμως η αρχή του πλήρους εναρμονισμού απέτυχε, τότε πρέπει κάποτε να φανταστούμε τι θα μπορούσε εναλλακτικά να λειτουργήσει. Και η ιδέα αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας είναι το εθελοντικού χαρακτήρα, προαιρετικού χαρακτήρα αυτό το μέσο. Στις διασυνοριακές συναλλαγές θα δημιουργήσουμε, είπαμε, μια δυνατότητα για τα συμβαλόμενα μέρη να ισχύει και να επιλέγεται ένα άλλο ε, συμβατικό πλαίσιο, ένα άλλο νομικό πλαίσιο που θα διαφέρει από τα εθνικά ε, καθεστώτα και θα είναι ένα ευρωπαϊκό δίκαιο συναλλαγών. Αυτή απομένει η ως τελική ε, επιλογή διότι αποκλείεται ο πλήρης εναρμονισμός. Και συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Τα γλωσσικά προβλήματα, τα πολιτισμικά και πολιτιστικά προβλήματα, οι διαφορές οι σημαντικά εμπόδια και προσκόμματα. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα εμπόδια και προσκόμματα δεν εμποδίζει και δεν παρακολεί κανέναν να μπορέσει να ακολουθήσει μια αναλλακτική λύση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και πράγματι, εδώ για τις διασυνοριακές συναλλαγές, θα, μια και δεν υπάρχει ε, ένα ενιαίο πλαίσιο, πρέπει αυτό να επιλεγεί για την προστασία τους. Και για μένα πάντα αυτός ήταν ένας λόγος. Γνώριζα ποιε είναι οι νομικές μας δυνατότητες και έτσι όταν θέλω να αγοράσω για παράδειγμα ένα έπιπλο, ε, για παράδειγμα εγώ από το Düsseldorf, να ε, μπορέσω να το αγοράσω εδώ ή ε, να μπορέσω να το αγοράσω αλλού σε σχέση με τη σύγκριση του κόστους. Διότι γνωρίζοντας ε, το ότι στην Ολλανδία έχουμε τις ίδιους, τους ίδιους όρους ε, για τις συναλλαγές αυτές, από πλευράς της πρακτικής του βιώματος ενός καταναλωτή επιλέγει κανείς τι κάνει. Επιλέγει κανείς από την πείρα του. Ένας συνάδελφος από το Λουξεμβούργο είπε πως το πρόβλημα από την πλευρά των προσφερόντων διαμορφώνεται και είναι γεγονός και το ξέρουν όλοι. Ο ή προσπαθούν στο διαδίκτυο να αγοράσουν κάποια προϊόντα και από, όταν προέρχονται από ένα μικρότερο κράτος μέλος. Πολύ συχνά αρνείται ο πάροχος και λέει ότι όχι δεν θα συμμετάσχω, δεν μπορώ να ε, συνεισφέρω. Οι εξετάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μελέτη επιπτώσεων ε, που καταδεικνύει ότι η εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ένας από τους λόγους για αυτή την κατάσταση είναι ότι ο πάροχος ε, δεν είναι δυνατόν και δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει παρατίθεται με κάθε ρύθμιση εθνικής νομοθεσίας στην Ευρώπη. Επιλέγουν λοιπόν τα, τις, τα πιο σημαντικά, τα ευρύτερα ε, ε, πλαίσια ε, νομολογίας μέσα στα οποία μπορούν να δράσουν και εγώ μπορώ να πω ότι η πρακτική ανάγκη είναι τεράστια να υπάρξει ένα τέτοιο μέσο διευκόλυνσης. Εδώ και πολλά χρόνια περιγράφεται αυτό. Όταν έχουμε ένα ακριβό αγαθό, ένα μεγάλων διαστάσεων ή μεγάλου αντιτίμου αγαθό που πωλείται διασυνοριακά, για παράδειγμα ένα μηχανικό εξοπλισμό, ένα κινητήρα, ένα μηχάνημα και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, εξεύρουμε μια δομή συμβατική που θα ανταποκρίνεται στις προσωπικές μας ανάγκες. Αν όμως είμαι ένας μικρός καταναλωτής ο οποίος ε, θέλει να αγοράσει ένα ε, εμπόρευμα 100, 150, 200 ευρώ διασυνοριακά από το διαδίκτυο με το παράδειγμα ενός ψυγείου για παράδειγμα ζω στην πόλη μου στο Düsseldorf θέλω να αγοράσω ένα ψυγείο από το διαδίκτυο βρίσκω κάποιον Ιρλανδό να το αγοράσω από αυτόν αυτό το ψυγείο. Και από έναν ε, Ρουμάνο μου παραδίδεται ένα τέτοιο ψυγείο. Έχω ένα τέτοιο ψυγείο το οποίο ίσως ε, κοστίζει 150 ευρώ και έχω μια τέτοια κατάσταση μπροστά μου. Ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί αν κάτι πάει στραβά. Το εθνικό μου δίκαιο το οποίο ισχύει στη Γερμανία. Το θέμα του πώς ε, μπορεί να ολοκληρωθεί μια τέτοια σύμβαση. Αν υπάρχουν ελλείψεις για παράδειγμα ή αν υπάρχει και ένα πρόβλημα μεταφοράς συνέχεια το ρουμανικό δίκαιο θα ισχύει σε σχέση με την μεταφορά αυτού του αγαθού. Και τώρα καταλήγω σε ένα δικηγόρο και λέω για την νομική μου κάλυψη νομικής ασφάλειας ε, θα ήθελα να αναλάβεις εσύ δικηγόρε αυτή την υπόθεση. Ε, δεν το πιστεύετε λοιπόν σας σοβαρά ότι αυτός ο συνάδελφος ο οποίος 50 ή 60 ευρώ θα πάρει θα κάσει και θα ασχοληθεί με το Ιρλανδικό δίκαιο, με το Ρουμανικό δίκαιο και στη συνέχεια θα μπορέσει να μου δώσει μια συνετή συμβουλή. Δεν θα πιστεύετε σοβαρά ότι ο αρμόδιος δικαστής ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει αυτό το θέμα στο Ντούσελ θα πάρει το Ιρλανδικό δίκαιο, το Γερμανικό δίκαιο, το Ρουμανικό δίκαιο, θα τα συγκρίνει και να δει τι θα πρέπει να εφαρμοστεί και πώ. Όταν έχει χιλιάδε τέτοιε περιπτώσει κάθε χρόνο. Και αυτό είναι αυτό το οποίο περιγράφηκε από πλευρά του καθηγητή πιο πριν, λοταρία. Είναι ένα είδο ε, κλήρωση αυτό. Δεν μπορούμε με τέτοια κλήρωση ε, θέματα τύχη και συγκυρία δηλαδή να ζούμε. Γι' αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των ε, δικαστών και των δικηγόρων στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και Συλλόγους των επαγγελματικών δηλαδή τη ε, ε, της επαγγελματικής εκπροσώπησης δικηγόρων για παράδειγμα είναι υπέρ αυτού του μέσου. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε λοιπόν να είναι ένα εύληπτο κατανοητό δίκαιο για όλους ώστε όλοι να μπορούν να κατανοήσουν περί πρόκειται. Αλλά εδώ έχουμε πράγματα τα οποία με πολλές εθνικές ρυθμίσεις ε, όπως ισχύουν αν δούμε τον αστικό κώδικα που ισχύει στη Γερμανία υπάρχουν παράγραφοι ολόκληρες, εδάφια ολόκληρα τα οποία έχουν συνταθεί από τον 19ο αιώνα και, έχουν συνε... Ε, ε, συνεχίζουν να υφίστανται και που κανένας δεν τα κατανοεί και είναι δυσνόητα για την πλειοψηφία των πολιτών. Και έτσι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα γεγονός λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθεί κανείς και να προβληματιστεί γι' αυτό και αυτό μπορεί να γίνει και με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής χωρίς καμιά αμφιβολία. Καταδείχθηκε ότι πρωτογενώ είναι ένα πρόβλημα του ηλεκτρονικού εμπορίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι μια απόλυτα καινούρια αγορά που δημιουργήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε και να πούμε ότι ακόμα και αν πρόκειται για τα πρώτα βήματα σε αυτή την εξέλιξη και νομοθετική ρύθμιση αυτού του τομέα αξίζει τον κόπο να ρυθμιστούν αυτέ οι πτυχέ Και μια τελευταία παρατήρηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, η δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων, model contract, ενός πρότυπου ε, ενός προτύπου σύμβασης. Όλα αυτά δεν υποκαθιστούν ένα τέτοιο λειτουργικό όργανο, διότι δεν επιλύουν τα προβλήματα τα οποία αναφύονται. Στο τέλος τέλος λοιπόν πρέπει να εγκρίνουμε μια πρόταση που θα δημιουργεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας καταναλωτών. Αυτό είναι και το αντίτιμο το οποίο θα πρέπει να δεχθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν να αντιμετωπίζουν 28 διαφορετικά νομικά καθεστώτα στην Ευρώπη, αλλά μόνο δύο, το εθνικό και για τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές ε, το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο διαμόρφωση συναλλαγών. Θα είναι λοιπόν ε, ένα δεδομένο πλαίσιο, δεν θα μπορεί κανείς ε, να επιλέγει εκείνο το οποίο ε, είναι μόνο το πιο επωφελές για αυτόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για όλους. Πάνω από το ελάχιστο επίπεδο το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί προστασίας καταναλωτών, βελτίωση σημαντική δηλαδή για την προστασία των καταναλωτών. Αυτά είχα να πω του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε θερμά αγαπητέ συνάδελφε Λένε. Μετά από την ε, σφαιρική διαφώτιση αυτή, φωτισμό των προβλημάτων, είναι φυσικά δύσκολο έτσι απλά να δώσει κανείς τον λόγο στη συνέχεια σε κάποιον άλλον, αλλά αυτό δεν ήταν η τελε, τελεσίδικη παρέμβαση, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Είναι σημαντικό το ότι για την πεμπτουσία αυτή των θεμάτων μας κάνετε να προβληματιστούμε. Σε αυτό θα ήθελα να δώσω τη σκητάλη τον λόγο στη συνέχεια λέγοντας δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να επικεντρωθούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο online εμπόριο, διαδικτυακά. Θα ακούσουμε το ένα ή άλλο σχόλιο ή παρατήρηση, όμως τον καθηγητή Σιμεωνίδη θα ήθελα πρώτα δώσω τον λόγο, να απαντήσει σε ερωτήσεις που διατυπώθηκαν ήδη. Παρακαλώ κύριε καθηγήτα. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ουσιαστικά ένα ερώτημα μου απευθύνατε. Θα προσπαθήσω, αν θέλετε βεβαίως, να απαντήσω και σε άλλα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ε, έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, όπως ο καθηγητής Μάιερ και είναι σε καλύτερη θέση να απαντήσουν. Πάντως, ε, ο γερουσιαστής από την Πολωνία μου έθεσε ένα ερώτημα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Γιατί να περιμένουμε, γιατί να γίνει τώρα αυτό. Ε, ε, ουσιαστικά εγώ το, τη χρονική διάσταση την έθεσα λίγο διαφορετικά. Σας ζήτησα να το ε, δείτε πιο μακροπρόθεσμα το θέμα της εναρμόνισης που, στην οποία μπορεί να μας οδηγήσει αυτό το νομοθέτημα εναρμόνιση οριζόντια σε θελούσια βάση και Εναρμόνες όχι μόνο για τις συνοριακές ε, αλλά και για εγχώριες. Αλλά δίκαιο έχετε που μιλήσατε και για την χρονική διάσταση ως ε, προς ε, τις κινήσεις της δικές μας. Δηλαδή πόσο χρόνο θα πρέπει να πάρει η επεξεργασία ενός τέτοιου νομοθετήματος. Ε, θα πρέπει ούτω ή να εργαστούμε καθημερινά για να βελτιώσουμε την πρόταση, αλλά είμαστε και ρεαλιστέ Είναι πελώριο αυτό το εγχείρημα και εξαιρετικά περίπλοκο. Εάν ακόμη και αν όλοι έκαναν το δικό τους κομμάτι της εργασίας, θα χρειαζόμασταν ε, χρόνο για να συζητηθεί το θέμα ε, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, γιατί έχουμε 27 κράτη-μέλη που ε, παρεμφερείς, αλλά και διαφορετικές νομικές παραδόσεις. Θέλουμε να εξετάσουμε μέχρι την τελευταία κυρία κάθε έγγραφο και από την εμπειρία μου, από τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας, δηλώνω ότι είναι απογοητευτικό ορισμένες φορές το αποτέλεσμα λόγω του χρόνου που παίρνει, αλλά δεν μπορούμε και να γίνουμε αντιπαραγωγικοί και να μην επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να ακούσουμε ε, τις ε, τοποθετήσεις όλων, ε, να σπέψουμε βραδέως δηλαδή, να ακούσουμε τις απόψεις όλων και να είναι καλό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αφήστε που δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, ενστάσεις, ε, αμφιβολίες, οπτικισμός όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλα βήματα που συζητείτε το θέμα. Τουλάχιστον τρεις ή και τέσσερις προεδρίες θα χρειαστεί το θέμα για να περάσει από το Συμβούλιο. Ίσως αυτό το χρόνο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε όλες οι υπόλοιπε ατέλειες. Πάντως χρειάζεται να συνεργαστούμε όλοι, δηλαδή το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όντω υπολείπεται μακρύ δρόμο, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξο και κυρίω να σκέφτομαι μακρόπνο και να διαβλέπω τα ενδυνάμει ωφέλη που θα απορρέουν από αυτό το εγχείρημα. Αυτό ήταν το μόνο ερώτημα νομίζω που μου απίφθηναν. Θέλετε μπορώ να προσπαθήσω να απαντήσω και σε άλλε, αλλά έχουμε εμπειρογνώμο εδώ, ο καθηγητή Θεάντερ Μάιερ που είναι ο εμπειρογνώμονα στο τομέα, νομίζω είναι σε καλύτερη θέση να απαντήσει. Ευχαριστώ ευχαριστούμε αυτό να κάνουμε τότε ε, για ο κύριος Σούλτεν ε, και νομίζω ε, θα πρέπει να απαντήσει σε δύο ερωτήματα. Μπορεί το κράτος, οι κρατικές αρχές να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συμβάσεις και δικονομικά ήταν η δεύτερη ερώτηση τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτο ερώτημα. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη συμβάση στο κράτο. Πρέπει να προσέξει κανεί σε ποια πλευρά θα παραμείνουμε. Στο ε, πρότυπο του e-commerce, ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι η καρδιά αυτών των συναλλαγών. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λόγο για του πελάτε, την πλευρά δηλαδή των αγοραστών. Η απάντηση τότε είναι όχι. Δεν μπορεί το κράτο να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδου συμβάσει εδώ σε σχέση με τους ε, καταναλωτές. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο δραματικό, διότι αυτό ισχύει για πολιτικά κόμματα, ιδρύματα ε, και αυτό τι σημαίνει πραγματικά στην πρακτική εφαρμογή. Ότι όπως έχει αυτή η διατύπωση ως σχέδιο αυτή τη στιγμή, οι επιχειρήσεις μόνο σε φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να πολλούν τα αγαθά τους. Όταν θα έχουμε ένα νομικό πρόσωπο από το εξωτερικό που θα παραγγέλει κάτι, θα πρέπει να διαπιστώνουμε αν είναι επιχείρηση ή μη επιχείρηση και σαφώς αυτό είναι δυσλειτουργικό και πρόκειται για μια αποδοχή χωρίς προβληματισμό των, ε, των ορίων της οδηγίας. Οδηγίες όμως ε, πληρούνται από τα κράτη. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοια συμμετοχή κρατών. Όταν λοιπόν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όταν προσεγγίζουμε αυτό το πεδίο, κάθε είδους ε, περιορισμός μπορεί να αρθεί το θέμα εδώ πρόκειται, ε, αφορά το θέμα των παρόχων και εκείνων που θα προσφέρουν τέτοια αγαθά. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ως πάροχοι ή ως προσφέροντες τα κράτη προβληματικό θα γίνει το πράγμα όταν αρχίζει κανείς ε, να έχει χρήστες ε, που θα πολλούν προς ε, άλλους χρήστες, καταναλωτές που θα πολλούν σε άλλους καταναλωτές. Εκεί πολλά θα μπορούσε κανείς πολιτικά να πει, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αναδιατυπωθεί τότε αν επιτρέπαμε όλου αυτού, όλες αυτές τις δυνατότητες. Δεύτερο, δικονομικά, ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο. Αυτό το θέμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απλό να απαντηθεί. Και ο πρόεδρος μας ήδη το προανέφερε. Είναι τυπικά το τοπικό τοπικά αρμόδιο ε, ε, δικαστήριο στην έδρα του χρήστη του καταναλωτή. Αυτό απορρέει από τις διατάξεις από τον κανονισμό ε, Βρυξελών 1. Νομίζω σε σχέση με το ιδανικό σενάριο δεν θα ήταν ε, ιδανικό αν πρωτογενώς ε, όλες τις αναπόφευκτες τριβές ε, τις οδηγούσαμε στα δικαστήρια. Στο ειρηνοδικείο για παράδειγμα στη Γαλλία, στο πρωτοδικείο για παράδειγμα στην Γερμανία είναι γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν ε, ε, για τα δικαστήρια να επιλαμβάνονται όλων αυτών των τριβών δεν θα ήταν καθόλου ελκυστικό κατέτιο για τους συμβαλόμενους. Ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό των ε, τριβών για παράδειγμα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε εξοδικαστικά να μπορεί να ρυθμίζεται και όσοι δεν θα ικανοποιούνται θα έπρεπε τότε να προσφεύγουν στα κρατικά δικαστήρια. Τελευταίο ερώτημα, το θέμα της αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Εξίσου αυτό και για το θέμα του, ε, της διευθέτησης των προβλημάτων στο ηλεκτρονικό ε, εμπόριο. Εδώ πραγματικά βλέπουμε ότι τα τοπικά δικαστήρια χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση ε, ε, δικαστών ε, να μπορούν να συγκρίνουν τις νομικές διατάξεις των κρατών μελών με ατέλειωτες διατάξεις και συγκρίσεις για να δουν μήπως αυτές θα ήταν καλύτερες ή χειρότερες σε σχέση με τις προβλεπόμενες. Εδώ πάρα πολλά μπορούν να απολεστούν διότι τα δικαστήρια σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους υπό 6.2 δεν μπορούν να εξετάσουν ε, σε αρκετό βάθος αν ε, οι επιλογές αυτές ε, είναι δεδομένες ή όχι. Το όλο αυτό σύστημα λοιπόν μόνο περιορισμένα μπορεί να λειτουργήσει. Είναι μια αποδοχή του σημερινού ε, ε, κράτους, του σημερινού καθεστώτος όπως λειτουργεί. Η απλή απλούστευση, η απλούστευση αυτών των διατάξεων μέσα σε ένα ενιαίο ε, πλαίσιο δικαιακά θα αποτελούσε ένα τεράστιο προτέρημα, ένα βήμα που θα βελτίωνε κατά πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Για το δεύτερο γύρο έχω τρεις που έχω ζητήσει τον λόγο συνάδελφος Νεράντζης Μαργαρέτα Σέντερφελτ και ο καθηγητής Στάουντενμάιερ. Με αυτή τη φορά, με αυτή τη σειρά θα πρότεινα να ακούσουμε τις παρεμβάσεις στη συνέχεια και πρώτα απ' όλα λοιπόν συνάδελφε Νεράντζη έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να υποβάλω ερωτήσεις με την άδειά σας. Μερικές ε, θέσεις θέλω να εκφράσω με πολύ δυνατή συντομία Καταρχήν χαίρομαι για το ότι εγκαταλείφθηκε πλήρω η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, μια εκδοχή την οποία είχα, στην οποία είχα αντιταχθεί στην περασμένη συνεδρίασή μας το 2010 εδώ στι Βρυξέλλε. Και επενώ το γεγονό ότι έρχεται η ρύθμιση με την πρόταση κανονισμού. Ε, παρά τα αυτά θέλω να διατυπώσω μερικές απόψεις. Πρώτον, η δημιουργία δύο παραλλήλων καθεστώτων με δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής δημιουργεί αναπόφευκτα ένα περίπλοκο σύστημα ρύθμισης των διαφορών επισυμβάσεων πώλησης το οποίο σύστημα ενδεχομένως να προκαλεί ασάφεια και ανασφάλεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύονται οι σχετικές διαφορές. Είδαμε ότι σε διαφορετικό μήκος κύματος αναφέρονται οι σχετικές παρατηρήσεις που ακούστηκαν προηγουμένως. Περαιτέρω, σε γενικό πλαίσιο και με εξαίρεση τη διάταξη του άρθρου 2 της πρότασης κανονισμού, όπου περιλαμβάνονται οι ορισμοί, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κρενόμενο κείμενο εκφεύγει από το τριμερές υπόδειγμα εργαλειοθήκη το οποίο είχε κατ' επανάληψη συμφωνηθεί στις συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων για κοινό δίκαιο της πώλησης, δηλαδή ορισμοί, αρχές, πρότυποι κανόνες. Καθώς επίσης και ότι τούτο διακρίνεται από ιδιαίτερο λεπτομεριακό χαρακτήρα σε αντίθεση με το χαρακτήρα λιτότητας και γενικότητας ο οποίος ομοίως άνω είχε συμφωνηθεί. Ε, ο καθηγητής κ. Βογγενάουερ έκανε μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις πάνω στο σημείο αυτό και για να δείξει ανάγλυφα τι έπρεπε να γίνει είπε σε ποιους άραγε απευθύνεται αυτό το κείμενο και προφανώς δεν εξέφραζε απορία ή δίλημα το κείμενο αναφέρεται σε εκείνους οι οποίοι ζητούν την προστασία σε εκείνους οι οποίοι, των οποίων οι σχέσεις ρυθμίζονται οι νομικοί παρεμβαίνουν αφήσει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι το κείμενο του προτινόμενου κανονισμού διασπά πολλαπλώς το δίκαιο της πώλησης. Ενδοσυνοριακές πωλήσει, διασυνοριακές πωλήσει μεταξύ καταναλωτών, C2C, μεταξύ επιχειρήσεων μικρής ή μεγάλης δυναμικότητας, B2B, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων C2B. Ειδικότερα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων προκύπτει ότι κάποια είδη της πώληση βάσει της υποδιαιρέσεως αυτής υπάγονται στο πεδίο του κανονισμού αυτού και άλλα δεν υπάγονται. Αφιβολίες περαιτέρω γεννώνται αναφορικά με το εάν αυτή η πολυδιάσπαση του δικαίου της πωλήσεως προάγει άραγε την ασφάλεια του δικαίου, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την κατοχυρωμένη καταρχήν ελευθερία των μερών να επιλέγουν ως εφαρμοστέο επί της συμβάσεως πώλησης που συνάπτουν όποιο δίκαιο επιθυμούν. Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ομοιομορφία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ρητή θέσπιση αριθμητικού ορίου σε ευρώ για τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Μιλάω για το άρθρο 7 του προτινομένου ε, κειμένου, καθώς η αγοραστική αξία του εν λόγου ποσού ποικίλει από χώρα σε χώρα, από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα και με τον πληθωρισμό. Τέλος, σημαντικό θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινιστεί κατά το σαφέστερο δυνατό τρόπο η σχέση του προτινόμενου κανονισμού με συναφή νομικά εργαλεία στα οποία τίθενται ζητήματα προστασίας του καταναλωτή. Ο κύριος Κιαοντόνε έθεσε προηγουμένως και επικαλέστηκε το θέμα της συμβάσεως της Βιέννης και είχε απόλυτα δίκιο. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ παράλληλα κείμενα κοινοτικά η οδηγία 29 του 2005 για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, η Οδηγία 31 του 2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας πληροφοριών και τον κανονισμό 539 του 2008, Ρώμη 1, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές ε, θα μπορούσα σε πολλά σημεία να διαφωνήσω με τις απόψεις του φίλου Προέδρου. Δεν έχω χρόνο καθόλου. Εκείνο που έχω να πω είναι μπορεί ένα νομοθέτημα να είναι παλιό, επικαλέστηκε τον Μπέγκεμπε, αλλά αυτή η παλαιότητα του κειμένου δημιουργεί ασφάλεια δικαίου. Και στις συναλλαγές τις ενοχικές, αυτές που αφορούν το δίκαιο της πολίσεως, η ασφάλεια δικαίου είναι το μείζον αγαθό. Ε, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με χαρά το κάναμε. Στη συνέχεια, Σέλαφελντ από τη Σουηδία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από σουηδικής πλευράς, πιστεύουμε ότι ο κανονισμός είναι και σημαντικός και απαραίτητος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των διασυνοριακών ε, συναλλαγών και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ταυτόχρονα βλέπουμε διάφορα διακριτά τμήματα στην πρόταση κανονισμού που θα πρέπει να μετεξελιχθούν και να διασαφινιστούν ούτως ώστε τα συμβαλόμενα μέρη να επιθυμήσουν να χρησιμοποιήσουν το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ε, διότι εάν δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τροποποιήσουν το νομοθέτημα θα φτάσουμε στο σημείο 0, στην αφετηρία. Για ποιο λόγο λοιπόν θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το νομοθέτημα τα συμβαλόμενα μέρη. Αυτό με φέρνει στις προτάσεις μας σε σχέση με τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν από ειδική πλευράς πάντοτε. Πρώτον, το επίπεδο. Δηλαδή, το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να δώσει μια ισορροπημένη προστασία των καταναλωτών στο ίδιο επίπεδο ανά την Ευρώπη και σε, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, τεχνικός πώς ε, να είναι εύχριστος ο κανονισμός και απλός στην εφαρμογή του είτε πρόκειται για συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις είτε για συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Δεύτερον, πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα των επιπτώσεων του κανονισμού. Δηλαδή θα πρέπει τα συμβαλόμενα να καταλάβουν ποιε είναι οι επιπτώσει, αν προκρίνουν αντίστοιχα το ε, οικείο, εθνικό δίκαιο ή αντίθετα το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με, με τη σωστή κατανόηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα συμβαλόμενα μέρη τι επίπτωσης ε, της εφαρμογής του ε, δικαίου. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι απλούστερη η διατύπωση. Τώρα, ε, στο νέο νομοθέτημα θα πρέπει να οριοθετήσουμε σωστά το περιεχόμενο, ούτω ώστε να γνωρίζουμε ποιες διατάξεις σχετίζονται με τις διασυνοριακές συναλλαγές. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να απαλληφθούν. Επίσης, ε, η νομική διατύπωση πρέπει να διευκρινιστεί, ούτω ώστε να είναι εύχριστος ο κανονισμός. Στη συνέχεια θα πρέπει η νομικός πως να είναι βιώσιμος ο κανονισμός, ε, δηλαδή να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σωστά σωστά. Τι εννοώ με αυτό. Ε, με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να εξετάσουμε ποια στοιχεία θα συμπεριλάβουμε, να δούμε πότε είναι εφαρμοστέο και πότε όχι το εθνικό δίκαιο. Μόνο όταν πληρούνται όλες αυτές ε, οι προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα της ενεργούς επιλογής ε, τα συμβαλόμενα μέρη και μόνο έτσι θα εφαρμοστεί το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλιώς εις προσπαθούμε να καταρτήσουμε ακούσουμε αυτό το νέο νομοθέτημα από ειδική πλευράς ε, δηλώνουμε πλήρη βούληση να συμμετάσχουμε στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και σε άλλα θεσμικά όργανα για αυτή την νομική πρόταση. Σα ευχαριστώ θερμά. Κύριε καθηγητά Μάιερ, πολλά θέματα αναφέρθηκαν. Για όλα τα θέματα μπορείτε να μας πείτε κάτι. Μας ενδιαφέρουν όλα, ιδιαίτερα σε δύο σημεία. Έχουμε ιδιαίτερη ζήτηση και ανάγκη. Ο μεγαλύτερος εστιασμός ε, στην, έτσι το ερμηνεύω εγώ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, online εμπόριο, μετά από τα όσα αναφέρθηκαν, αλλά και για τα θέματα του 114 άρθρου της ε, συνθήκης και σε σχέση και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς από πλευρά της Επιτροπής θα θεωρούν τα πράγματα και σε όλα τα άλλα θέματα. Σας δίνω τον λόγο να τοποθετηθείτε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τέσσερις παρατηρήσεις θα κάνω μόνο και θα προσπαθήσω να απαντήσω και στα δύο δικά σας ερωτήματα. Το πρώτο σημείο που προέρχεται από τον Λόρδο Μπάουνες και τον Σερ Άλαν Στον πρώτο γύρο των συζητήσεων αναφέρθηκαν εκεί δύο στο θέμα των τεκμηρίων που ζητάει η Βρετανική κυβέρνηση αληθεύει αυτό. Έλαβαν 40 τέσσερις συνεισφορές, εκ των οποίων 23 ήρθαν από ενώσεις ε, καταναλωτών ε, και επαγγελματιών του κλάδου. Όλες ήταν αρνητικές. Οι 43 συνεισφορές προήλθαν από ε, φυσικά πρόσωπα, από ακαδημαϊκούς, από συλλόγους, ενώσεις, μεμονωμένους δικηγόρους, από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό είναι και το πρώτο στοιχείο της απάντησής μου. Δύο ε, θέσεις ε, μας ήρθαν από ε, συλλογές επιχειρήσεων αυτές οι δύο ενώσεις εκπροσωπούν σχεδόν ολόκληρο το λιανικό εμπόριο, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Και οι δύο θέσεις ήταν θετικές. Γιατί? Εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να σας παραβέψω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ε, οι περισσότεροι καταναλωτές σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζουν επιγραμμικά. Οπότε οι δύο αυτές ε, ενώσει που εκπροσωπούν όπω σα είπα σχεδόν το σύνολο του λιανικού εμπορίου ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να εκμεταλλευτούν ακόμη περισσότερο αυτή τη δυνατότητα και άρα επιθυμούν να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο ε, εν είδη απάντηση. Το δεύτερο, το, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Ελενέ, ε, η τρεις νομικές υπηρεσίες επικύρωσαν την επιλογή του άρθρου 114 για νομική βάση, αλλά αν κοιτάξει κανείς ε, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, σε σχέση με το άρθρο 114 και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για νομικές ε, προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι ίσως υπάρχουν συγκεκριμένοι φράγμοι για το εμπόριο αλλά πρέπει να καταδειχθεί αυτό. Ε, δεν είναι δύσκολο να το στοιχειοθετήσουμε. Αν δούμε συμβάσει, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσει καταναλωτέ, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσει, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ εθνικέ ε, υποχρεωτικέ ε, διατάξει. Τώρα, μπορεί να καλύπτονται και τομείς ε, όπου ε, δεν εφαρμόζεται ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά υπάρχουν ε, αποκλίνουσες οικίες εθνικές διατάξεις. Αυτό συνιστά νομικό πρόσκομα. Στη συνέχεια, η μελέτη αντικτύπωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξε ότι αυτές οι διαφορές συνεπάγονται και οικονομικό κόστος. Υπολογίσαμε ότι για μια φυσιολογική επιχείρηση για να εξάγει σε μία και μόνο χώρα... Ε, απαιτούνται 10.000 ε, ε, ευρώ και 3.000 ευρώ αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ιστοσελίδα. Άρα υπερβαίνεται ουσιαστικά το ετήσιο τζίρο μιας μικρής επιχείρησης εν τη αυτή περιπτώσει. Δηλαδή μπορεί να είναι απαγορευτικό το κόστος ε, και πολλοί συναλλασσόμενοι ε, δεν εξάγουν ή επιλέγουν μόνο ένα ή δύο κράτη-μέλη προς τα οποία θα εξάγουν. Το ίδιο κόστος ε, ισχύει και για τις συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αποδείξαμε ότι υπάρχουν νομικά και οικονομικά προσκόμματα για τις συμβάσεις επιχειρήσεων προς καταναλωτές αλλά και για ε, τις συμβάσεις επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις. Οπότε το άρθρο 114 ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση και αυτή είναι ε, η αιτιολογία που επιλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο που, ε, ζήτημα που γύρε ο κύριος Ελένε για την επικουρική νομική βάση του τεστ είναι το άρθρο 352. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο και αυτό παγιώνεται μέσα στην ομολογία του 10, μόνο εάν το άρθρο 114 δεν είναι ε, ε, δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση και εμείς προτείναμε ε, λύση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή έχουμε διαμορφώσει το πεδίο εφαρμογή με τέτοιο τρόπο, δηλαδή συμβάσεις όπου εμπλέκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ανταποκριθούν στις ε, δικές μας απαιτήσεις. Ε, δεν καλύπτουμε χωρίς πωλήσει, δεν καλύπτουμε συμβάσεις ανάμεσα σε μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί εκεί δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα. Άρα διαμορφώσαμε αναλόγω το πεδίο εφαρμογή. Ε, τώρα, η δυνατότητα χρήση επικουρική νομική βάση του άρθρου 352. Σα αποδείξω γιατί δεν γίνεται, αλλά ακόμη και αν το εξετάσουμε ω υποθετικό σενάριο. Υπάρχει και σχετική νομολογία για εμπορικά σήματα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται ε, για τα ίδια ζητήματα. Δηλαδή, όταν ε, μιλάμε για την υπόθεση παραδείγματο χάρη εμπορικών σημάτων, ε, για την οποία απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, παραδείγματο χάρη, η δεύτερη υπόθεση του ΔΕΚ, δεν ε, είναι μια νέα νομική εντότητα. Δηλαδή, δεν μεταφέρεται αυτή η εταιρεία σε ένα άλλο κράτο μέλο, απλώ δίνεται η δυνατότητα ε, να μεταφερθεί η ίδια εταιρεία χωρίς να δημιουργηθεί νέα νομική εντότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά σήματα. Σε αυτή την περίπτωση η δημιουργία νέων νομικών οντοτήτων ε, ε, μπορεί να προβλεφθεί μόνο από τους νομοθέτες. Ε, αυτό τι σημαίνει, αν χρησιμοποιήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό δίκαιο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 352 όμως εμείς ε, εδώ πραγματευόμαστε ένα εντελώς ε, διαφορετικό ζήτημα. Δηλαδή δεν δημιουργούμε μία νέα νομική οντότητα ούτε μία νέα μορφή σύμβασης. Έχουμε μία σύμβαση και δύο συμβαλόμενα μέρη που μπορούν ε, με πλήρη αυτονομία να επιλέξουν ένα σετ κανόνων και να δημιουργήσουν μία δική τους σύμβαση ε, που διέπεται κανονικά από το εφαρμοστέο, δηλαδή το εθνικό δίκαιο και έχουν την δυνατότητα στα πλαίσια του οικείου εθνικού δικαίου να προκρίνουν ένα εναλλακτικό ε, νομικό σύστημα. Αυτό είναι εντελώς, ε, μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Το άρθρο 352, ακόμη και ως επικουρική νομική βάση, δεν είναι εφαρμόστεο σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό με φέρνει στο σημείο που σχολίασε ο κύριος Κρίγκερ, δηλαδή την επιλογή του καταναλωτή. Πιστεύω ότι υπάρχει μια παρανόηση από πλευρά ε, σα ε, σχετικά με το ανακοινωθέν ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι ο, ότι ο καταναλωτή θα έχει την επιλογή ανάμεσα στο οικείο εθνικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το έχει. Ο έμπορος, ο πολιτής μπορεί για την διασυνοριακή αυτή συναλλαγή να έχει αυτή την επιλογή και να επιλέξει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οπότε ποια επιλογή υπολείπεται για τον ε, καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να μην αγοράσει αυτό το προϊόν ε, και να ε, πάει στο κατάστημα κάτω στη γωνία γιατί ξέρει ότι είχε μόνο θετικές εμπειρίες, δηλαδή είχε πρόβλημα, το πήγε πίσω στο κατάστημα το προϊόν, το επέστρεψαν στην επιχείρηση και το ξαναπήρε επιδιορθωμένο. Ε, ή όταν υπάρχει κάποιο ελότημα, ελάττωμα, συγγνώμη, ο καταναλωτής ε, θέλει να μπορεί να μιλήσει με κάποιον και μπορεί να ε, προτιμήσει να πληρώσει 10% παραπάνω, αλλά να πάει στο κατάστημα της γειτονιάς, γιατί είναι σημαντικό για αυτόν να έχει ένα συνομιλητή. Μπορεί επίσης επιγραμμικά να αγοράσει κατά 10% φθηνότερα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Εξαρτάται αν είναι σημαντική η οταν υπαρχει καποιο ελοτημα ελαττωμα συγγνωμη ο καταναλωτης θελει να μπορει να μιλησει με καποιον και μπορει να προτιμησει να πληρωσει 10 παραπανω αλλα να παει στο καταστημα τη γειτονιά, γιατι ειναι σημαντικο για αυτον να εχει ενα συνομιλητη μπορει επίση επιγραμμικα να αγορασει κατα 10 φθηνοτερα βασει του ευρωπαικου δικαιου εξαρταται αν ειναι σημαντικη η τιμη για τον καταναλωτή. Μπορεί να το κάνει αυτό γιατί μπορεί να πρόκειται για ένα αγαθό με συγκεκριμένη εμπορική η ονομασία στο οποίο έχει εμπιστοσύνη και γι' αυτό είναι αυτό πιο σημαντικό και την έχει την επιλογή ο καταναλωτής. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευρύτερη επιλογή με το νέο σύστημα ο καταναλωτής, κάτι που δεν διαθέτει τώρα και έχει πιο ανταγωνιστικές, φτηνότερες δηλαδή μέσα; αλλά και πάλι διατηρεί την επιλογή να πάει σε ένα κατάστημα ε, κοντά στον τόπο διαμονής του. Αλλά αυτό δεν επαρκεί. Όταν ο καταναλωτής επιλέξει το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο, μπορεί τελικά να καταλήξει ε, σε μια χειρότερη θέση από ότι αν ε, είχε εφαρμοστεί το εθνικό δίκαιο. Δύο εμπειρογνώμες μας το είπαν αυτό ήδη σήμερα, δηλαδή ένα κοινό δίκαιο πολίσεων ε, ε, προσφέρει μία προστασία, επίπεδο προστασίας καταναλωτών ίσο ή ανώτερο σε σχέση με όλα τα εθνικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και δεύτερον προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας υψηλότερο από τα επίπεδα που κατοχυρώνονται βάσει των εθνικών δικαίων. Δηλαδή μπορεί να επιλέξει να αγοράσει ε, ευθυνότερα προϊόντα αλλά και από νομικής πλευράς είναι καλύτερα προστατευμένος ο καταναλωτής. Δεν μπορεί να χάσει δηλαδή βάση του νέου συστήματος. Του προσφέρουμε μια επιλογή που δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή γιατί τώρα ο πολιτής μόνο μπορεί να επιλέξει το εφαρμοστέο δίκαιο και αν δείτε το άρθρο 62 του κανονισμού Ρώμη να μπορεί να επιλέξει μόνο το εθνικό δίκαιο. Και εμείς του προσφέρουμε τώρα ένα δίκαιο που είναι ίσο ή καλύτερο από το εθνικό δίκαιο. Από νομικής πλευρά λοιπόν αποκλείεται να βγει χαμένος και έχει και τα οικονομικά ωφέλη επιπροσθέτως. Αυτή ήταν η τρίτη παρατήρησή μου. Η τέταρτη παρατήρηση τώρα για να απαντήσω στις ερωτήσεις που άκουσα εδώ. Ε, και βάσει της μελέτης του καθηγητή Φόγγενάουερ και βάσει των δηλώσεων ε, του κυρίου Λένε σε σχέση με τις αδυναμίες ως προς τη διατύπωση του νομικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με τα σχόλια του Λόρδου Μπάνουσε και τη τα σχόλια του Προέδρου για τις επιγραμμικές ε, αγορές. Θα ήθελα όλα αυτά να τα ομαδοποιήσω και να σας πω τα εξή. Πρώτον, ο καθηγητής Φόργεν είπε κάτι που βρίσκω ενδιαφέρον. Είπε ότι το, η φρασιολογία του ευρωπαϊκού δικαίου είναι καλή συμβαστική λύση ανάμεσα σε διάφορα ε, στυλ διατύπωσης ε, που υπάρχουν στην Ευρώπη. Έτσι μας είπε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό έτσι, ε, αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Ε, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το στυλ διατύπωση γιατί πάντοτε έχουμε το δίλημα ανάμεσα στην ευελιξία και τα πράγματα που πρέπει να καλύψουμε. Εμεί θέλουμε τον κοινό παρονομαστή. Αυτό επιλέξαμε και το επιβεβαίωσε και ο καθηγητή. Ε, και τώρα επανέρχομαι στι ατέλειε σε σχέση με την διατύπωση και εδώ θα ήθελα να παραθέσω κάτι στα γερμανικά γιατί πρόκειται για μια δήλωση που έγινε στα γερμανικά. Ελπίζω όμω ότι μέσα τη μετάφραση να κατανοήσετε το συνέστημα και τη συναισθηματική φόρτιση. Ξεκινώ το παράθεμα. Έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί η υπόθεση. Αλλά τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει τώρα. Από τότε που διατυπώνεται αυτό το ερώτημα, η γραμματολογία, η βιβλιογραφία έχει πάρει διαστάσεις ολόκληρης βιβλιοθήκης πια πολυάριθμες και αξιοπρόσεκτες προτάσεις για βελτίωση στα επιμέρου τμήματα του σχεδίου αναφύονται και προτάθηκαν. Εν μέρη σοβαρές φωνές ακούστηκαν με προτάσεις για την περαιτέρω εκπόνηση του νομοθετικού αυτού εγχειρήματος. Κανείς, κανείς από ό,τι μπορούμε να αξιολογήσουμε δεν ήταν υπέρ της ε, χωρίς, τροποποιημένες, ε, χωρίς έγκριση αυτού του σχεδίου. Θα μπορούσα να σας αφήσω να μαντέψετε ποιος το είπε αυτό. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια τέτοια, ένα τέτοιο παράθεμα θα μπορούσε από τη συζήτηση αυτή να προέρχεται ήταν ο Otto von Γκιόκεν και αυτό έγινε το 1889 στην Γερμανία σε 30 χρόνια εκπονήθηκε μετά από 30 χρόνια ο κώδικας αστικού δικαίου. 112 ολόκληρα χρόνια ε, λειτουργήσε και η εκτίμηση ήταν ότι ήταν αρκετά καλός ε, και από πλευράς διατύπωσης. Δηλαδή νομοθετικά ο νόμος μπορεί να βελτιωθεί στη διατύπωσή του, στην εκδοτική διατύπωση και ουσιαστικά και εδώ επανέρχομαι σε αυτό το οποίο ανέφερε ο καθηγητής Σιμεωνίδης στις δύο συναντήσεις στο Συμβούλιο υπό την Κυπριακή Προεδρία είχαμε αρκετές καλές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από, το, από τα κράτη-μέλη για τη διατύπωση του κεφαλαίου 10 και αυτό συζητήσαμε και υπήρξαν βελτιώσεις και θα συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση, αυτή η πορεία και ευελπιστώ προ αυτό. Ουσιαστικά σε μια μεταγενέστερη φάση μπορούμε να έρθουμε και στο θέμα του φάσματος, του εύρους και πάλι εδώ σε σχέση με τις ε, συζητήσεις για περιορισμούς ε, που σε αυτή τη φάση όμως είναι πρώιμη η συζήτηση. Πρώτα πρέπει να συζητήσουμε την ουσία προτού περάσουμε στο εύρο στην εμβέλεια. Εδώ όμω σε μια τέτοια πρόταση μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να πούμε ότι και μια τέτοια πρόταση όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί, να τύχει βελτιώσεων. Και αυτό το οποίο είπε και ο καθηγητής Σιμεωνίδη. Ας βελτιωθούν λοιπόν αυτά από το Συμβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θερμά, ε, σας ε, ευχαριστούμε θερμά καθηγητά ε, Μάιρ για τα όσα μα είπατε. Εδώ έχουμε αφενό την ανάγκη να καταλήξουμε σε ένα ε, ευρωπαϊκό ε, κοινό πλαίσιο δικαίου όσον αφορά τις συναλλαγές, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο online. Έχουμε όμως και πολλά ερωτήματα τα οποία ανεφίσαν που πρέπει να τα επεξεργαστούμε για να τα απαντήσουμε. Και αν κατάλαβα καλά τα πώς αυτά που είπατε κύριε καθηγητά Στάουντενμαϊερ που αναφερθήκατε στον γερμανικό αστικό κώδικα στα, στους πέντε τόμους ε, και Γνωρίζω και από την ε, ε, γενέθλια πόλη ότι έχουμε και μια δεύτερη επιτροπή που εργάστηκε μετά στη συνέχεια μέχρι γύρω στο 1900 να μπορέσει να εγκριθεί η διατύπωση από πλευράς του νομοθετήματος. Διερωτώ με πώς μπορούμε να καταφέρουμε το στόχο που θέλουμε να ευδοκιμήσει και να στεφθεί με επιτυχία και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ αυτά, αλλά έχω τον εισηγητή δίπλα μου. για αυτό, αυτό το τομεακό θέμα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον ε, ε, κύριο Λένε. Ευχαριστώ θερμά καθηγητά και ευχαριστώ και για το ότι εσείς αναλάβατε το ρόλο του συντονισμού και το ότι μπορέσατε να συντονίσετε με εξαιρετικό τρόπο το δεύτερο πάνελ. Είναι δύσκολο μια και κατέληξε στα συμπεράσματά του ο καθηγητής υποβάλλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο νομοθέτης εγκρίνει. Νομοθέτης είναι το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ούτε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την νομοθετική διαδικασία δεν απέρευσε όπως προτάθηκε. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι η ανάγκη της ε, σε εξέλιξη διαδικασίας work in progress στα αγγλικά έργο ή εν ρευστό ε, εν εξελίξη και για τους, ε, τους προβληματισμούς μας πώς αυτό το νομοθετικό έργο μπορεί να βελτιωθεί στο τέλος είμαστε ευγνώμονες για όλες τις προτάσεις προτάσεις που προέρχονται από τους πραγματογνώμονες τους επαΐοντες από τα Εθνικά Κοινοβούλια θερμά ευπρόσδεκτες είναι, καλοδεχούμενες πρόγραμμά μας είναι να υπάρξει ένα έγγραφο εργασίας των δύο εισηγητών το έχετε νομίζω ε, στα χέρια σας και η πρόθεσή μας είναι αυτό το έγγραφο εργασίας κατά την αρχή του, ε, της Άνοιξης ε, γύρω στο, στα τέλη Φεβρουαρίου-Μάρτιο να έχουμε ένα, μια πρώτη, ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσής μας όπου θα ανοιχνεύσετε, θα ανοιχνεύονται κάποιες τάσεις και κατευθύνσεις να αναλύσουμε τα προβλήματα τα οποία απορρέουν και από την ακρόαση και με όλα τα έγγραφα τα οποία καλύψαμε προτείνοντας δημιουργία γεωργικές ευφυείς λύσεις. Μετά θα ακολουθήσει μια υστερότερη φάση της άτυπης διατύπωσης ε, με τους συμβαλόμενους, τους εμπλεκόμενους, όλους τους ενδιαφερόμενους και μετά από πρώτες συζητήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου, την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, θα δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το εγχείρημα, ποια συνέχεια θα δοθεί στη συνέχεια σε συνεργασία με τους δύο συνομοθέτες ε, που συμμετέχουν ε, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θέλω να σας πω ότι σαφέστατα είναι η πρόθεσή μας στην Ευρωβουλή με ιδιαίτερη ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα να προσεγγίσουμε το νομοθετικό αυτό έργο. Στόχος μας είναι στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό έργο που θα στεφθεί με επιτυχία. Δεν θέλουμε θνησιγενές δίκαιο, θέλουμε ένα λειτουργικό, ζωντανό δίκαιο, το οποίο θα είναι θελκτικό, ελκυστικό, χρήσιμο, λειτουργικό. Και γι' αυτό α, χρειαζόμαστε τον αναγκαίο χρόνο για να τα κάνουμε όλα σωστά. Αναφερθήκατε στο χρόνο που απαιτήθηκε ώστε το εθνικό αυτό έργο, νομοθετικό έργο να καταλήξει στον εθνικό Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα. Δεν θα χρειαστούμε εμεί τόσα πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι περιοριζόμαστε μόνο σε κάποιε συγκεκριμένε ε, πτυχέ ε, συμβάσεων συναλλαγών αγοραπολισιών. Άρα λοιπόν είναι σαφέστερο το πλαίσιο και πιο περιορισμένο. Όμω, ε, εδώ σε σχέση με τα όσα έγιναν κατά τη δεκαετία του 80 σε σχέση με τις, ε, τα όσα προετοιμάστηκαν προλιάθηκε το έδαφος κατά τη δεκαετία του 1990. Επί δεκαετίες έχουμε προχωρήσει. Φτάσαμε τώρα σε μια χρονική συγκυρία όπου ορίμασαν τα, ορίμασε η χρονική συγκυρία ώστε να καταλήξουμε σε ένα σωστό θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να σας προαναγγείλω ότι η Νομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου πριν από λίγες μέρες πρόσφατα αποφάσισε ότι του χρόνου το 2013 θα διεξαγάγουμε μια τέτοια συνδιάσκεψη σαν αυτή που είχαμε σήμερα κατά το δεύτερο εξάμεινο και πάλι ώστε να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις και τα θα έχουν απορρεύσει σε αυτή τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μαζί σας δηλαδή κυρίες και κύριοι. Και να συνεχίσουμε με μια δεύτερη ακρόαση. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αμοιβαία μας εμπλουτίζει με την ανταλλαγή επιχειρημάτων επί τη ουσία και προτάσεων, προτάσεων πώς αυτό το προϊόν για το οποίο κάνουμε λόγο μπορεί ακόμα περαιτέρω να βελτιωθεί. Σα ευχαριστώ θέρμα, ευχαριστώ όλου που ήρθατε και συμμετείχατε σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Τώρα, ολοκληρώνοντας, σας προσκαλώ να πάμε για ένα ποτό σε μια δεξίωση. Δεξίωση στο κτίριο, μια στιγμή να δω, Γιάν Γιώζε Αντάλ κτίριο, εδώ δίπλα, είναι το κτίριο που περνάτε την Πασαρέλα, τη γέφυρα και μετά πάτε λοξά αριστερά στο τέλος του διαδρόμου. Οι συνεργάτες της γραμματείας θα σας βοηθήσουν να βρείτε εκεί το σημείο. Θα παραμείνουμε στον ίδιο όροφο, δεν χρειάζεται να πάρετε ανελκυστήρα, να πάρετε ασανσέρ, να μετακινηθείτε αλλού. Θα χαιρόμουν να έβρισκα τον έναν ή άλλον από εσά και να ξανασυζητούσαμε κάποια θέματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ για τις προτάσεις και τα επιχειρήματά σας και την υποστήριξη. Γεια!